Bene. Bentrovati a tutti. Buonasera a tutti. Καλησπέρα σε όλους.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε συζητήσει επανειλημμένως τη σημασία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την σύμφωνη γνώμη του για τον κανονισμό του Συμβουλίου για το πολιετές πλαίσιο, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει και είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας να εργαστεί επί νομοθετικών προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής σε στενή συνεργασία με τους του Επιτροπή Προπολογισμού που φέρουν την ευθύνη για την δημοσιονομική διαδικασία του πολιτού πλαισίου. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχής και ευγνώμων που οι συνάδελφοι Ράιμερ Μπόγκε και η Βάιλ Κάλφιν μέσως και, και πρόθυμα δέχτηκαν την πρόσκλησή μας για μια ανταλλαγή απόψεων για τα διαδικαστικά θέματα. Θα μας ενημερώσουν επίσης και τους ευχαριστώ και γι' αυτό για την ε, κατάσταση προόδου στην Επιτροπή Προπολογισμού και για την ε, διαδικασία που θα ακολουθηθεί ώστε να συζητήσουμε τη συμμετοχή των ειδικευμένων επιτροπών, των κυριολεκτικών επιτροπών και φυσικά εμείς είμαστε μια επιτροπή που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ε, κατάσταση προόδου των εργασιών ε, για το σε πλαίσιο και για τις προβλέψεις που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Ευχαριστώ βεβαίως και τον εισηγητή Τζαν Κάρλο Σκοτά που είναι εισηγητής για τη γνωμοδότηση αλλά θα αρχίσουμε δίνοντας το λόγο καταρχήν στον κύριο Ράιμερ Μπέγκε που θα μας ενημερώσει. Παρακαλώ Ράιμερ, έχεις το λόγο. vielen Dank, ευχαριστώ. Χαίρομαι που είχα, έχω την ευκαιρία και πάλι να έρθω στην Επιτροπή και θα ήθελα να σημειώσω ότι θα πρέπει να μοιραστούμε με τον γιατί το, την παρουσίαση. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, την συναπόφαση, 65 με 70 πολιετή προγράμματα δηλαδή και σε μια νέα εποχή θα έλεγα των πολιτικών διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να διαφυλάξει την παράλληλη έκβαση, το συντονισμό δηλαδή των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και, που είναι και αρμοδιότητα της Επιτροπής των Προϋπολογισμών και των πολιετών προγραμμάτων που θα πρέπει να ε, προχωρήσουν κατά τρόπο ορθολογικό. Ξέρετε ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο μόνο εφόσον έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη με πλειοψηφία των μελών του το Κοινοβούλιο πρώτα. Στο θέμα λοιπόν αυτό της συναπόφασης, η συνέλευση, σταγματική συνέλευση στο τέλος των διαδικασιών της, των εργασιών της, ε, ε, ε, έγινε μαλλιά κουβάρια για να το πω απλά και περιληπτικά στο άρθρο 312.5 παράγραφος 5 ορίζεται ότι θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να προσδιορίσουν κατά τρόπο λογικό, ορθολογικό τι διαδικασίε του να μπορούν να προχωρήσουν διαδικασίε και η λήψη αποφάσεων χωρί προβλήματα. Οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ε, ω προ το συντονισμό και ω προ την ε, εξασφάλιση μια επιτυχού έκβαση για τη διαδικασία. Και έτσι στην υλοποίηση της συμφωνίας η οποία είχε, η συναυθεί με την Ουγγρική ε, Προεδρία άρχισε να εφαρμόζεται στην Πολωνική Προεδρία και τώρα συνεχίζεται υπό την Δανική. Γίνεται μια συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιο για το δημοσιονομικό πλαίσιο, με προσδορισμό, με παρουσίαση μάλλον τη πραγματευτική του Συμβουλίου ε, στο τρίο του, στην τριανδρία του Συμβουλίου για να ενημερώσει και να ενημερωθεί για τις ε, εξελίξεις στην, ε, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Έχουμε μια Έχουμε μια πενταμελή ομάδα που εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο ε, με τον κύριο Λαμασούρ, τον Ιβανο Κάλφιν, τον υποφαινόμενο και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου Μάρτιν Σούλτς και με συμμετοχή βεβαίω όλων των ε, συντονιστών από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ήσασταν και εσεί παρόντες πιστεύω στην παρουσίαση της ομάδας επαφής του Κοινοβουλίου και τη συζήτηση στην οποία λάβατε μέρος για την, ε, τις διαπραγματεύσεις. Η οριστική διαδικασία πιστεύω θα ε, συζητηθεί και θα εγκριθεί οριστικά πλέον από διάσκεψη των Προέδρων σύντομα. Είχαμε μια συζήτηση για το πώς ε, θα χειριστούμε το θέμα από εδώ και μπρος, αν θα κάνουν οι επιτροπές την προετοιμασία για την πρώτη ανάγνωση, αν θα κάνουμε την ψηφοφορία για το τελικό κείμενο. Αλλά όταν δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα, ποια είναι τα ποσά, συγκεκριμένα ποσά, δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για μεταρρυθμίσεις, για τροποποιήσει, ε, για τροπολογίε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινό στα θεσμικά όργανα. Και ε, σημαντικό αυτή τη στιγμή θεωρώ το ότι μου φαίνεται αδύνατον με να προσδιοριστούν ε, ε, για τα πολιετή προγράμματα συγκεκριμένα ποσά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως πρόγραμμα για την Επιτροπή ΣΟΥΡ, την προσωρινή δηλαδή Επιτροπή, όπου είπαμε ότι τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, αυτό που προβλέπει και η Λισαβόνα, αυτό που ορίζει και η Ατζέντα 2020. Είπαμε 20 συν 30% συν 2% από πληθωρισμό μέχρι ότου υπάρχουν οριστικά στοιχεία, οριστικές αποφάσεις σε άλλο επίπεδο. Και ταυτόχρονα ορίσαμε μέσα από την ε, συνθήκη ότι σε περίπτωση όπου δεν θα εξασφαλιστεί συμφωνία τα ανώτατα επίπεδα για τον ε, προϋπολογισμό του 2013 θα ισχύσουν και θα επαναλαμβάνονται τα ανώτατα επίπεδα κάθε χρόνο μέχρι ότου εξασφαλιστεί συμφωνία σε επίπεδο πολυετών ε, του δημοσιονομικού πλαισίου. Και σε αυτό, Πρόεδρε, με κάπως προκλητικό τρόπο, θα έλεγα ότι απλά το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να συζητά, χρειάζεται απλώς να αναπαυθεί και να περιμένει να προχωρήσει το Συμβούλιο σε κάποιες ε, υποχωρήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπει σε ένα παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε, πρέπει να διαπραγματευτούμε δηλαδή. Η ιδανική προεδρία έχει ξεκινήσει με τα λεγόμενα negotiation boxes, τα ε, διαπραγματευτικά κοιτία, που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες και όπου συζητείται το πόσο θα χειριστούμε αυτά τα διαπραγματευτικά κοιτία, δηλαδή αν μπορούμε να επισέλθουμε εις βάθος, αν μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για ποσά, πλαίσια, προτάσεις, περαιτέρω διαβούλευσης. Η Προεδρία της Δανίας κλήθηκε από μας να δώσει το ταχύτερο δυνατό ε, στοιχεία, να μας δώσει έγγραφα, τεκμηρίωση για να μπορούμε να κρίνουμε τις ε, προτάσεις της και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι και η Επιτροπή των Προϋπολογισμών αλλά και οι επιμέρους επιτροπές πρέπει εγκαίρως με να κάνουν τη δουλειά τους αλλά και να μιλήσει μόνο ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα πριν να συμφωνηθούν τα πάντα και ότι εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα ε, δεν ικανοποιηθούν αιτήματα συγκεκριμένα για έναν τομέα καταρρύπτεται ολόκληρη, πίπτη μάλλον ολόκληρη η συμφωνία ε, όσον αφορά το Κοινοβούλιο. Εν πάση εμεί ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια κάποια πρόοδο. Είμαστε σε αναμονή του Συμβουλίου του Ιουνίου, ίσως του Ιουλίου, που πιστεύουμε ότι θα αντιδράσει. Μια ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής των Προϋπολογισμών ε, μπορεί να κατατεθεί αρχάς Οκτωβρίου και στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων πιστεύω θα έχουν ε, την δυνατότητα και οι επιμέρους επιτροπές, οι, οι ειδικευμένες επιτροπές να δώσουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτές είναι οι συνθήκες πλαισίου για μένα. Ο κύριος Κάλφιν, συνεισηγητής, ίσως έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήταν σαφέστατο ο κύριο Μπέγκε. Ίσως καλύτερα να ακούσω πρώτα τις ερωτήσεις και να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις τεθούν. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπέγκη και τον συνάδελφο Κάλφιν ακόμα μια φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνάδελφε Φι, αυτά που μας είπαν. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω το θέμα της έκθεσης Γαρίγα, αυτή που εμείς εγκρίναμε στην Ειδική Επίτροπη ΣΟΥΡ. Για μας αυτό αντιπροσωπεύει την πρόταση του Κοινοβουλίου και σαφώς όλες οι ομάδες είναι προσανατολισμένες στην υπεράσπιση αυτής της έκθεσης που, είχε, που έλαβε τεράστια πλειοψηφία όχι μόνο στην Επιτροπή ΣΟΥΡ αλλά και στην Ολομέλεια και το Θυμίζω και διευκρινίζεται αυτό πολύ ξεκάθαρα Η ε, στόχη εκεί του Κοινοβουλίου. Τώρα το Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις του. Εμείς ήδη ε, δώσαμε τη γνωμοδότησή μας και είναι πολύ σημαντικό επίσης και ε, θα ήθελα να το υπογραμμίσω ακόμη μια φορά δεν έχει αποφασιστεί μέχρι ότου να έχουν αποφασιστεί όλα. Το ακούσαμε αυτή τη φράση πολλές φορές και στην συνεδρίαση της ομάδας επαφής και είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την επιχειρηματολογία του Κοινοβουλίου. Έχουμε πολλούς ε, που θέλουν να μιλήσουν, αλλά εγώ θα ξεκινήσω με τον Τζαν Κάρλο Σκοτά, βεβαίως, που είναι ο εισηγητής μας υπεύθυνο για την σύνταξη της νομοδότησής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους δύο τεχνικούς ε, συναδέλφους της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Οι προκλήσεις που μας περιμένουν και οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής μας υποχρεώνουν να έχουμε συμπαγή θέση μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής μας, μέσα στο πλαίσιο του συζήτηση για το πολιετές πλαίσιο, γιατί εκεί έγκυται το μέλλον των ε, γεωργών μας. Τα σενάρια που, εξετάζονται μέσα στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου είναι τρία και από αυτόν θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Η πρόταση, η είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αξίες που, χρησιμοποιεί, που προτείνει. Χρησιμοποιεί ως βάση αναφορά στα νούμερα του 2011. Ο αριθμός για τη δεύτερη κατηγορία ε, και που σχετίζεται με την βιώσιμη ανάπτυξη τους ε, φυσικούς πόρους είναι περίπου 380 δις ευρώ. Σημαίνει αυτό μείωση του 7% σε σχέση με το προηγούμενο πολιετές πλαίσιο. Στη συνέχεια είναι το πρόταση της Επιτροπής ΣΟΥΡ και είναι αυτή της γενικής αύξησης 5% ε, σε σχέση με τον προπολογισμό του 2013 με εκείνο το 2% που μόλις ακούσαμε. Ο προπολογισμό του 2013 που θα έχει παγώσει σύμφωνα με τις τιμές του 2011 και θα ανέρχεται περίπου στα 410 δις ευρώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και εδώ έχω αναφέρει νούμερα αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νούμερα παρά μόνο μέχρι ότου να ξέρουμε τελικά ποια θα προταθούν και τι θα έχουμε στη διάθεσή μα. Το τρίτο σενάριο είναι η διατήρηση του status quo στο επίπεδο του πολιετού πλαισίου του 2007 με 2013 που αν υπολογίσουμε μια ετήσια έναν ετήσιο υποπληθωρισμό φτάνει στα 420 δις ευρώ. Εάν λάβουμε υπόψη το άρθρο 312 της συνθήκης που λέει ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου που ορίζει νέο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν εγκριθεί ε, μέσα στην ε, προβλεπόμενη προθεσμία, παρατείνονται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το προηγούμενο έτος μέχρι ότου ληφθεί απόφαση. Δηλαδή αυτό θα είναι το σενάριο που μας περιμένει εάν δεν υπάρξει απόφαση. Ο προπολογισμό του 2013 και βεβαίως με έντονη συνεργασία μπορεί εμείς να καταφέρουμε και να σημάνουμε τη διαφορά για τους ε, γεωργούς μας. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας φυσικά και θα ακούσω προσεκτικά όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε Τζαν Κάρλο Σκοτά και ξεκινάμε τη συζήτηση με τον George Λάιον. Ε, thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλη αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας διότι υπάρχουν διάφορα δημοσιονομικά ζητήματα που θα κυριαρχήσουν ή ήδη κυριαρχούν στις συζητήσεις μας. Αν συμφωνήσουμε με την διαδικασία αυτή, όπου η ομάδα επαφής και οι συγητές διαπραγματεύονται, τότε θα πρέπει να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη για να τα καταφέρουμε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Ρένχαρτ Μπόγκε για το σημείο κίνησης και όλα αυτά, γιατί αυτά έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον ε, γεωργικό προπολογισμό. Υπάρχουν ε, μερικά ζωτικά ζητήματα για την Επιτροπή Γεωργίας. Πρώτα απ' όλα, στο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την αναβολή της αύξησης του 4,5% για την περίοδο 2007-2013, το πάγωμα δεν είναι σε πραγματικούς όρους. Οπότε Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Δεύτερον, η μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή μας ήταν το θέμα της ανακατανομής των απευθείας των άμεσων πληρωμών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα. Και θα είναι δύσκολο να πιστούν τα μέλη της Επιτροπής μας να το δεχτούν. Θα πρέπει οι απόψεις μας να περάσουν στο έγγραφο εργασίας. χρειάζεται να μας καθισχάσουν οι εκπρόσωποι εδώ της Επιτροπής Προϋπολογισμών για να μπορέσουμε να τους εμπιστευτούμε στη συνέχεια. Πρέπει να μας καθησυχάσουν για το τι θα γίνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να ξαναδούμε τις νομοθετικές διατάξεις και τις προτάσεις που έχουμε ήδη ψηφίσει για να δούμε τελικά ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Όλη αυτή η διαδικασία βασίζεται στη διαφάνεια, στο ανοιχτό πνεύμα. Αλλιώς θα βρεθεί ο ένας τομέας να μάχεται τον άλλον. Από πλευράς πάντως Επιτροπής Γεωργίας πρέπει να προσέξουμε πολύ και να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και να δούμε αν ε, θελήσει το Κοινοβούλιο να απορρίψει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Το πάγωμα είναι καλύτερη στάση από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να το ζυγίσουμε πάρα πολύ καλά πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Τέλος, επειδή είμαι μέλος της ε, ομάδας επαφής, θα κοιτάξω και αυτά τα συμφέροντα βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Όντω πρέπει να κάνουμε ομαδικό παιχνίδι. Ο κ. Σόσλινγκ και μετά ο Μισελ Νταντά. ναι, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι που έχουμε. Μπορούμε να είμαστε ευτυχεί που έχουμε τον Ράινερ Μπέγκε ε, στο πιδάλιο. και με βέβαιο ότι έχουμε ισχυρά επιχειρήματα στην υπόθεση αυτή, αλλά από την άλλη ό,τι και να λέμε δεν μπορούμε να θεωρούμε και να στοιχηματίζουμε ότι θα είμαστε καλύτερη κατάσταση αν παγώσουν οι προπολογισμοί. Μόνο κατάσταση ανάγκη μπορεί να μα οδηγήσει στον αποτέλεσμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμω για τι διαπραγματεύσει, μια ερώτηση για τον Ράιναρ Μπέργκερ. Πώ βλέπει τα πράγματα. Τι προβλέπεις. Γιατί μπορεί πάντα να λέμε ότι υπάρχουν κρατημέλη τα οποία θέλουν να επιβάλλουν πολύ σημαντικέ περικοπέ και να λέμε ότι. ενώ οι κάποιοι άλλοι να λένε ότι δεν θα πληγεί από κάποιε περικοπέ ο προπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, εάν είναι σοβαρέ οι περικοπέ, προφανώ και θα πληγεί και ο προπολογισμό για τη γεωργία από τι περικοπέ αυτέ. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφέ, να το εξηγήσουμε. Η δε ανακατανομή των ποσών, πράγμα που συστήσαμε και παλαιότερα, είχαμε και μια αντιπροσωπεία από κράτη της Βαλτικής που είχαν εκδηλώσει την δυσφορία τους για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ε, προβεί σε τόσο διαφορετικές πληρωμές, καταβολές ποσών δηλαδή για τον πρώτο πυλώνα και τώρα βλέπουμε ότι μπορεί η ε, αναδιανομή των ποσών να οδηγήσει σε πολύ επώδυνες ε, περικοπές. Για δε το χρονοδιάγραμμα βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής που πρέπει να είναι φιλόδοξη, χωρίς όμως να ξέρουμε πόσα χρήματα θα έχουμε στη θέση μας για να την υλοποιήσουμε. Πιστεύω ωστόσο πάντα και το συζητούμε και συχνά στην Επιτροπή μας ότι πρέπει να διατυπώσουμε μια πολιτική γεωργική με μια πολιτική γεωργική ορθολογική ώστε να είμαστε σε θέση και να προβάλλουμε την ε, σοβαρότητα της δουλειά που θα έχουμε κάνει και όταν θα έχουμε τα ποσά, έστω και αν δεν έχουμε τώρα ποσά. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά για τον εξορθολογισμό της γεωργικής πολιτικής Και βέβαια για την υλοποίηση θα πρέπει να, είμαστε, να βρούμε μια συμφωνία μας το 2013. Ευχαριστούμε. Ο Μισελ Νταντά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ ε, τα δύο μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που ήρθαν να ανταλλάξουν μαζί μας απόψεις. Το είπαμε ήδη ότι το Κοινοβούλιο εκφράστηκε με σαφήνεια. Στην Επιτροπή μα ήμασταν ορισμένοι εκεί, στην Επιτροπή αυτή, εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας και ε, στις εργασίες που έγιναν εκεί και ακούσαμε και μας άκουσαν. Για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχουμε ως στόχο το να καταλήξουμε κάπου μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής, ή τέλος πάντων το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2013. Αλλιώς, ολόκληρη η εικόνα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πλήττεται, ζημιώνεται. Και δεν μιλώ μόνο για τη γεωργία και το γεωργικό προπολογισμό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογέ το 2014. Αν λοιπόν αρχές του 2013 δεν είμαστε σε θέση να καθορίσουμε προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πάρα πολύ δύσκολο λίγου μήνε αργότερα θα πάμε μπροστά στο εκλογικό σώμα για να υποστηρίξουμε τι θέσει μα. Εγώ είμαι εισηγητής για το τμήμα που αφορά τη ΣΚΟΑ τις κοινέ οργανώσεις αγοράς. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τους δύο συναδέλφους. Στην δημοσιονομική πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Κομισιόν υπάρχει ένα γεωργικό προπολογισμό. Υπάρχουν χρήματα τα οποία απευθύνονται στην γεωργία ε, από το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν ε, κονδύλια για τη διαχείριση της κρίσης που αμφισβητούν άλλοι. Αλλά έτσι κι αλλιώς και στη και στην άλλη περίπτωση για να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά υπάρχουν μακρές και περίπλοκες διαδικασίες. Πιστεύετε λοιπόν τώρα που προβληματιζόμαστε και πάλι για τους δημοσιονομικούς ε, μηχανισμούς που θα ισχύσουν στην επόμενη περίοδο, μήπως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα μας ε, πέτρεπε να κρατάμε τα πλεονάσματα από τον γεωργικό προϋπολογισμό και να τα μετακινούμε. Δηλαδή τι εννοώ, αυτά τα πλεονάσματα μπορούμε να τα κρατήσουμε για τρία χρόνια, τότε μπορούμε σε περίπτωση κρίσης να έχουμε έτοιμα τα χρήματα για να παρέμβουμε και αν δεν υπάρχει κρίση, τότε επιστρέφουν στα κράτη-μέλη τα χρήματα αυτά όπως κάναμε και μέχρι τώρα. Με ένα τέτοιο σύστημα το οποίο βέβαια είναι μια παρέκκληση από τα όσα ίσχυαν μέχρι τώρα, ένα τέτοιο σύστημα θα είχε σαν αποτέλεσμα να ε, προσφέρει κάποια ασφάλεια στον γεωργικό ε, προϋπολογισμό και θα επέτρεπε να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά όταν πραγματικά χρειάζονταν. Ο καιρός που πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε θέμα κρίσης και ότι έτσι κι αλλιώς η αγορά θα τα όλα, έχει τελειώσει ο καιρός ε, αυτός. Το καταλάβαμε νομίζω και από χτες το απόγευμα από αυτά που είπαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση λοιπόν, να μπορούμε δηλαδή κάτι να κάνουμε και για να μπορούμε κάτι να κάνουμε πρέπει να έχουμε χρήματα. Εγώ δεν λέω να φτιάχνουμε θέματα, λέω όταν υπάρχουν πλεονάσματα από τη διαφορά στη τιμή. Αν μη τι άλλο, έτσι μπορούμε να καλύψουμε την παραγωγή και να καλύψουμε και την κατάσταση σε περίπτωση κρίσης. Ελένη και μετά Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική συζήτηση αυτή που κάνουμε και ευχαριστώ τους συναδέρφους από την Επιτροπή προεπολογισμών που ήρθαν να μας παρουσιάσουν τις κύριες ιδέες όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τα πράγματα. Ο συντονισμός λοιπόν ακριβώς αυτός θα εξαρτηθεί ή τέλο πάντων ανάποδα να το πω, η κοινή γεωργική πολιτική θα εξαρτηθεί από τον καλό συντονισμό που θα κάνουμε εδώ, γιατί χρειαζόμαστε φυσικά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χρειαζόμαστε και έναν μεγάλο προπολογισμό, γιατί έχουμε ένα σωρό προγράμματα. Θέλουμε το πρασίνισμα της ε, ΚΑΠ, θέλουμε τους μηχανισμούς παρέμβασης ε, της αγοράς. Ένα σωρό πράγματα που θέλουμε απαιτούν περισσότερα χρήματα. Πρέπει λοιπόν αυτές τις πληρωμές να τις δούμε ισορροπημένα, γιατί η κατάσταση είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Όλα αυτά έχουν ένα τίμημα. Φυσικά και ο χρόνος παίζει ρόλο. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε στο Κοινοβούλιο, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Όλοι λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γνωρίζουμε και εγώ βέβαια που είμαι και μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή, γνωρίζουμε λοιπόν ότι άπαξ και υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των διαφόρων τομέων, αυτό θα ήταν καταστροφικό για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει δηλαδή να μπούμε σε ανταγωνισμό μεταξύ μας και ο καθένας να λέει το δικό του, ένας να λέει α, περισσότερα στην ανάπτυξη, περισσότερα στη γεωργία, ο άλλος και ούτω καθεξής. Όχι. Πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ μας και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν και αυτά γρήγορα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χρειαζόμαστε πολιτικέ για την απασχόληση, χρειαζόμαστε πολιτικέ για την ανάπτυξη και για το περιβάλλον. Και θέλουμε επίση και η Γεωργία να μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω εσεί στην Επιτροπή Προπολογισμών πώ το βλέπετε αυτό. Εμεί πάντως Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει και να μας παρουσιάσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που όλοι χρειαζόμαστε και αυτό να το κάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να μπούμε στις διαπραγματεύσεις έχοντας επίγνωση των συνεπειών. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον που στην Επιτροπή μας. Η μεταρρύθμιση Πάντοτε λέω, είναι όπω το hardware και το software, το υλικό και το λογισμικό. το λογισμικό το κάνουμε εμεί, το υλικό εσεί, από την Επιτροπή των Προπολογισμών μα εξασφαλίσετε τα κονδύλια για να την υλοποιήσουμε. Και τότε μόνο θα μπορούσαμε βεβαίω να ε, συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε σε αποφάσει για τη μεταρρύθμιση τη γεωργική πολιτική τότε και μόνο τότε όταν θα έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία δεδομένα ποσά για τον προπολογισμό. ίσως μέχρι και τελευταία στιγμή να παίζουμε πόκερ στην υπόθεση αυτή, δεν ξέρω. Ε, μερικά ερωτηματικά. Πρώτον, από τα κράτη-μέλη πόσα χρήματα εισραίων. Λέτε, υπάρχει μια πρόταση επιτροπής. Πολύ καλά. Η γερμανική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει λίγο πολύ ότι θα διαθέτει 1% επί του ΑΕΠ της Γερμανίας ως συμβολή με κοινοβουλευτικές διαδικασίες ε, διαφορετικά. Εάν θέλει να ξεπεράσει λέει, το 1% πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της κοινοβουλευτικής έγκρισης. Είναι καλό αυτό το 1%. Καλή είδηση, κακή είδηση. Μας φτάνει, αντέχουμε, χρειαζόμαστε κι άλλα. Καταστροφή, τι απ' όλα. Δεύτερον, αποπληθωριστής, deflator. Είναι ένα είδος ε, αποθεματικού στον προϋπολογισμό. Καλό να υπάρχει, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Η Επιτροπή πάντως είχε προετοιμάσει διαφορετικές εκδοχές σχεδίων του προϋπολογισμού. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχετε αντιληφθεί πως ξεκαθάρισε η εικόνα και εάν έχει ποσοστό σε αυτόν τον αποπληθωρητή η γεωργική πολιτική ή όχι. Τρίτη ερώτηση. Η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση η οποία προφανώς επηρεάζει και το ΕΠ μπορεί να επηρεάσει τις ε, Ε, επηρεάζει μήπως τα απόλυτα ποσά του ΑΕΠ και ως εκ τούτου και τα ποσά των εισφορών στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω αν υπάρχει δυνατότητα να δούμε ένα χαρτί, ένα έγγραφο στο οποίο να δούμε ξεκάθαρα την εικόνα, την περίπτωση Φερρυπίν τη μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει πολύ μεγάλη επιστροφή από τι εισφορέ στον προπολογισμό, Εν μεταξύ έχουν βρει και άλλοι τον δρόμο τη επιστροφή, αρκετά σημαντική. Αλλά πάση το χρονοδιάγραμμα πώς το προβλέπετε εσείς. Ε, ποια θα ήταν μια ρεαλιστική προσέγγιση. Πότε μπορούμε να περιμένουμε να δούμε έναν προπολογισμό πάνω στον οποίο να, να μπορούμε πραγματικά να δουλέψουμε εγκαίρως και όχι πολύ αργά. Ευχαριστώ πολύ Μπρίτα μας και μετά Ζεμποβέ. Κυρία Ρέινας, πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στους ε, εισηγητές, εισηγητές. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Και ξεκάθαρα ακούστηκε ότι το Κοινοβούλιο μπόρεσε με την έκθεση Σούρε να προσφέρει σημαντική συμβολή στην υπόθεση αυτή. Τώρα πρέπει το Συμβούλιο να κάνει τις ορθολογικές του προτάσεις, να ανταποκριθεί δηλαδή στην προσφορά τη δική μας. Βέβαια, εμένα ως ε, γεωργό με ενδιαφέρει το, όχι μόνο το να γνωρίζουμε τι είδους ποσά μπορώ να εργαστώ. Αλλά βάσει τίνος επίας ε, γεωργικής μεταρρύθμισης μπορώ να εργαστώ για να ξέρω και τι ποσά θα υπάρχουν αλλά και πώς μπορεί ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος να προγραμματίσει τη δουλειά του γιατί ξέρετε ότι αυτή εξαρτάται πάρα πολύ από τις αλλαγέ των εποχών και τις συγκεκριμένε εποχές του χρόνου και άρα πρέπει να είναι στη θέση εγκαίρως να φυτέψουν τη μία ε, σοδιά ή την άλλη. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να επιδείξουμε πνεύμα Σοβαρότητα, Απαιτούμε να έχουμε την ενημέρωση εγκαίρω και επαρκώ, σε επαρκή βαθμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταλήξει σε απόλυτες προτάσεις ο προπολογισμό, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση λίγο πολύ. Ξέρουμε πόσο ε, τραβάνεις μάκρος οι διαπραγματεύσει. Ξέρουμε πόσο τραβάει μάκρο η διαδικασία σε επίπεδο διοίκηση, πόσο χρόνο χρειάζεται η διοίκηση για να υλοποιήσει τι προτάσει. Και μόνο αφού καταφέρει η διοίκηση να θέσει σε εφαρμογή τι προτάσει, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι υλοποιούνται τα μέτρα. Ε, και όταν ήρθε αυτή τη στιγμή, πια ο Γεωργό έχει χάσει το τρένο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον. Και άρα νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα περισσότερο έναντι του Γεωργού του κτηνοτρόφου και λιγότερο του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το, το διακύβευμα εδώ. Επίση, πολύ σημαντικό είναι Εάν έχουμε ένα πρότυπο νη συν 6, αν ακολουθούμε ένα πρότυπο νη συν 6 και πούμε ότι ε, ισχύουν, εξακολουθούν να ισχύουν τα κονδύλα του προπολογισμού. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο όμω ότι το έχουμε λύσει το πρόβλημα, γιατί έχουμε ένα προπολογισμό τη γεωργική πολιτική, ο οποίο τρέχει ακόμη. Έχουμε μια γεωργική πολιτική που τρέχει ακόμα, που όμω έχει χρονικά όρια και πρέπει να αναλάβουμε μέτρα κατά τρόπον υπεύθυνο και ορθολογικό για την πολιτική. Για την ύπεθρο, τι θα κάνουμε δηλαδή με όλα τα προγράμματα υποστήριξη για την ε, για το δεύτερο πυλώνα, Φερρυπίν πώς θα βρούμε τις ε, φάσεις ε, για τα επόμενα προγράμματα και τα έργα που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει και δεν είναι γνωστά. Βλέπω λοιπόν ότι έχει τεράστιες ευθύνες στο Συμβούλιο και έχει τεράστιες ευθύνες στο Συμβούλιο για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο και πρέπει να ε, αναλάβει τις ευθύνες του και να ε, ικανοποιήσει τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται ε, επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν ξέρουν τι θα πράξουν την επαύριον. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι έχει έρθει πια η ώρα να ληφθούν οι αποφάσεις, να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να επιφορτίζεται με την ε, λήψη απόφασης ή να ε, χρεώνεται μία αποτυχία το Κοινοβούλιο, όταν το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο δεν έχει θεωρήσει πως ακόμα έχει έρθει η ώρα να ε, ξεκινήσει τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις. Εμείς η Επιτροπή ε, για τα γεωργικά θέματα πρέπει οπωσδήποτε όλη αυτή τη συζήτηση να την προβάλλουμε και στην κοινή γνώμη, να ενημερωθεί ο κόσμος, να γνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει, ότι το Κοινοβούλιο κόπτεται να προχωρήσει, αλλά το Συμβούλιο είναι αυτό που ψέρνει τα πόδια του. Ευχαριστώ σας, Και μετά Μαγκίνες. Euh, Ακούω τη συζήτηση αυτή που γίνεται για τον προπολογισμό και νομίζω ότι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Προπολογισμών κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν μια ορθή θέση, οικονομικά ορθή θέση. Το πρόβλημα όμως δεν το έχουν αυτοί, το έχουμε εμείς, Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσο δεν έχουμε καθορίσει το τι θέλουμε, τι δηλαδή γεωργική πολιτική θέλουμε, δεν θα έχουμε κανένα συγκεκριμένο μέσο για να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας για έναν προπολογισμό. Σήμερα δουλεύουμε ανάποδα. Αν ξεκινάμε μόνο από το ότι θέλουμε να διατηρήσουμε έναν προπολογισμό, αυτή είναι η αρχή μας, και μετά ανάλογα με τα χρήματα που θα έχουμε, μετά θα βάλουμε το τι θέλουμε να κάνουμε, μετά δηλαδή θα ταιριάξουμε την πολιτική μας στα χρήματα που έχουμε, ε, τότε δεν θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάτι σωστό. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε ένα πραγματικά πολιτικό πρόβλημα εδώ στο Κοινοβούλιο μας και στην Επιτροπή αυτή Γεωργίας. Πρέπει να καθορίσουμε πρώτα απ' όλα τη γεωργία που θέλουμε και μετά αυτό να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε με τον κατάλληλο προπολογισμό, το ανάποδο, δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά. Δεν γίνεται. Κάνουμε την ανάπολη δουλειά από αυτή που θέλουμε. Είτε πρόκειται λοιπόν για το πρασίνισμα, είτε πρόκειται για το περιβάλλον γενικότερα, είτε πρόκειται για τη στήριξη των ε, γεωργών απέναντι σε μια κρίση. Χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Αλλά τι βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε σήμερα ότι το σχέδιό μας είναι κατακαιρματισμένο, ότι δεν υπάρχει τίποτα εγκάρσιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα απέναντι στις άλλες επιτροπές. Γιατί σήμερα είμαστε μέσα ε, σε μια κρυστάλλινη γυάλα. Και όσο είμαστε εκεί μέσα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και μπορεί να θέλουμε ε, να συμφωνήσουμε με τις δύο πολιτικές μεγάλες ομάδες, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έτσι είναι σαν να μένουμε στο περιθώριο και να προσπαθούμε έτσι να ψιλοκανονίσουμε τα πράγματα, να τα διευθετήσουμε. Όχι, αν θέλουμε ε, γεργούς, αν θέλουμε προϊόντα που να συνδέονται με τη γη όπου παράγονται. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, δεν θα τα καταφέρουμε με από τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε Μάλλον να μην δεχτούμε να συζητήσουμε για έναν όγκο χρημάτων αν δεν έχουμε πρώτα την πολιτική μας, γιατί δεν είναι τα χρήματα που θα μας δώσουν την πολιτική μας, αλλά το ανάποδο. να ακούσουμε την ε, απάντηση του και την αντίδραση του Ράιμερ Ντελάγκε. Συγγνώμη που δεν έδωσα προηγουμένω το λόγο. Η κυρία Ντελάγκε είναι εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά δεν το είχα καταλάβει κι εγώ. Άκουσα όμως ε, τον κύριο Ποβέ και εδώ μας βάζει ένα συνδυσιακό πρόβλημα. Όντως, θα έχουμε διαφορά μεταξύ μας για το τι πολιτική θέλουμε για τη γεωργία. Συμφωνώ όμως με αυτό που λέτε για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ότι δηλαδή η δικιά μας η δουλειά, αυτό που πρέπει εμείς ε, να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα που λέει γιατί η γεωργική πολιτική παίρνει το 35% του προπολογισμού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Δύο πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ευρωπαϊκή πολιτική, άλλο είναι το ότι γίνεται σε εθνικό επίπεδο, εντάξει, σωστό. Αλλά στην πολιτική συζήτηση καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν παίζουν και πολύ σημασία. Το δεύτερο είναι να φροντίσουμε για την ασφάλεια τροφίμων πολύ σωστό. Είναι ο πυρήνα και πρέπει να παραμείνει να είναι ο πυρήνα τη γεωργική μα πολιτική η ασφάλεια τροφίμων. Αυτό είναι που πρέπει ε, να πούμε και να εξηγήσουμε γιατί θέλουμε το 35%. Αυτή είναι η δικιά μας η δουλειά λοιπόν. Αυτό να εξηγήσουμε. Να δείξουμε ποια είναι η στρατηγική σημασία που έχουν τα τρόφιμα και γιατί θέλουμε αυτό το ποσοστό από τον ε, Ευρωπαϊκό Κορβανά. Τώρα η σημερινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πράσινο, το ξέρουν και οι συνάδελφοι, ότι για μένα είναι κάτι που δεν θα λειτουργήσει. Εγώ θα το ήθελα διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε πέρα από τα τρόφιμα, γιατί άλλο έχουμε τη γεωργία, τι άλλη κοινωνική χρησιμότητα έχει η γεωργία πέρα από την παραγωγή τροφίμων να μιλήσουμε για τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, να συζητήσουμε για ε, φωσφορικά και άλλες ε, ουσίες που χρησιμοποιούνται. Τέτοια πράγματα να πούμε και να δείξουμε ότι η γεωργία δεν είναι μόνο για τους γεωργούς. Βέβαια είναι καταρχήν για τους γεωργούς. Οι γεωργοί φυσικά και πρέπει να κερδίζουν το ψωμί τους με την ε, δραστηριότητά τους. Αλλά η γεωργία δεν είναι μόνο για τους γεωργούς, είναι για την κοινωνία ολόκληρη. Τότε έχουμε μια καλή ιστορία που μπορούμε να παρουσιάσουμε και να δικαιολογήσουμε τα χρήματα που ζητάμε. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει εμείς να κάνουμε, να βρούμε δηλαδή τα σωστά επιχειρήματα και αυτό πρέπει να το κάνουμε και γρήγορα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε κυρία Ντελάγκη και τώρα η Μαρίν Μακίνες και μετά ο Λαβία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολλές ερωτήσεις που ήθελα εγώ να έχω απαντήσεις ε, τις υπέβαλε ο Πίτερ Ευχαριστώ λοιπόν Πίτερ και ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, του προπολογισμού. Εγώ θα ήθελα ίσως ε, κάποιες προβλέψεις. Ξέρουμε ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου που είναι ξεκάθαρη, αλλά από τα διάφορα μηνύματα που μας έρχονται από το Συμβούλιο δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς σημαίνουν. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε κάπως. Και έπειτα, πώς λειτουργεί η συναπόφαση όταν οι επικεφαλείς ε, κρατών πάνε σε μια αίθουσα και συμφωνούν για τα σημαντικά νούμερα. Εμείς σε αυτή τη δικασία πού βρισκόμαστε, έξω από την πόρτα, ακούμε από το παράθυρο, πώς λειτουργεί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε. Και αν το Κοινοβούλιο θέλει να σταθεί στο ύψο του και δεν είναι ικανοποιημένο με τον προπολογισμό, μπορεί να πει όχι, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα. Θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική που σημαίνει ότι αν πούμε όχι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το τι θα κάνουμε μετά, τι θα ακολουθήσει. Τι θα γίνει, θα είμαστε σε καλύτερη θέση. Ποιες θα είναι οι συνέπειες σε τέτοια περίπτωση. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για αυτή τη διαδικασία, γιατί κατά κάποιο τρόπο είμαστε μπλοκαρισμένοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ή δεν θα εξελιχθούν μέχρι το τέλος του έτους. Και με τις διάφορες επιλογές που θα γίνουν μέσα στους επόμενους 24 μήνες, πώς θα επηρεάσουν όλα αυτά τον προπολογισμό. Ευχαριστούμε Μάριαντ. Ο Τζοβάνι Λαβία και μετά θα ξαναπάρει το λόγο η προσκεκλημένη μας. Ε, εγώ περισσότερο εδώ μιλώ ως ε, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και, αλλά και ε, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας γιατί είμαι κάπως ανάμεσα στις δύο επιτροπές. Αλλά κάτι που είναι προφανές από την αρχή ε, της συζήτησης που κάναμε για αυτό το επόμενο πολιετές πλαίσιο είναι ότι οι προτάσεις που προέρχονταν για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής είχαν συνταχθεί για να υπερασπιστούν τον προϋπολογισμό που, είχε, που προοριζόταν για την κοινή πολιτική. Η νομοθετική πρόταση δηλαδή που μας υπέβαλε η Κομισιόν είναι μια νομοθετική πρόταση ε, έτσι φτιαγμένη ώστε να είναι δυνατόν να υπερασπιστεί τον προπολογισμό που προορίζεται για την κοινή πολιτική και αυτό πρέπει να είναι σαφές για όλους. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για τα οποία είμαστε μπερδεμένοι στη συζήτηση εδώ σε αυτή την Επιτροπή και μιλώ για το πρασίνισμα κυρίως, αλλά και για άλλα μέτρα και άλλες παρεμβάσεις, αυτό οφείλεται στο ότι στο εσωτερικό της συζήτηση για το πολιετές πλαίσιο χρειάζεται να έχουμε συμμάχους, χρειάζεται να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης ε, γιατί έτσι ώστε να συνεχίσουν να προορίζονται σε αυτές τις πολιτικές ένα, ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θεωρώ πως είναι σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι η νέα γεωργική πολιτική δεν μπορεί να απαντά μόνο στις παλιές προκλήσεις όπως έλεγε για κάποιος που μίλησε προηγουμένως. Είναι απαραίτητο και συγκεκριμένα να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις που απαιτούν φυσικά μια συνεπή ε, δέσμευση των πόρων. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω άλλη μια φορά ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν ΣΟΥΡ, δηλαδή του, για το πάγωμα και όχι πάγωμα προς τα κάτω όπως προτείνει η Κομισιόν αλλά πάγωμα του γεωρικού προπολογισμού του 2013 ε, αυτή είναι η πρόταση που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε και να στηρίξουμε με ε, δύναμη με Σε Ευχαριστώ Τζοβάνι. Ας ακούσουμε τις απαντήσεις του κυρίου Καλφίν και φυσικά μετά αν ο Μπέγκε θέλει να παρέμβει θα μπορέσει. Σας ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω και ο κύριος Μπέγκε θα συνεχίσει και θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Αρκετές ε, ομάδες ερωτήσεων έχουμε. Καταρχήν, Νομίζω πως η ουσιαστική ερώτηση την οποία έθιξε ο κύριος Μποβέ παραμένει. Δεν θα πρέπει να συζητάμε μόνο νούμερα ή το επόμενο πολιτές ε, πρόγραμμα θα πρέπει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για πολιτικές. Συμφωνώ σε αυτό και αυτό είναι ένας ε, από τους λόγους για τους οποίους ήθελα να πάω σε όλες τις επιτροπές και την Γεωργική Επιτροπή στις συνομιλίες με το Συμβούλιο ακριβώς έτσι ώστε να τεθεί το θέμα των πολιτικών. Διότι Όλοι είμαστε ρεαλιστέ εδώ, δεν αναμένουμε θαύματα όσον αφορά την χρηματοδότηση. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα όπως και στους εθνικούς προπολογισμού, ενώ ταυτόχρονα έχουμε πολύ ψηλότερες φιλοδοξίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποια μικροποσά εδώ και εκεί ή αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε πολιτικέ. Εάν δούμε τι προτάσει τη επιτροπή, υπάρχουν κάποιοι τομεί όπου δεν υπάρχουν αλλαγές πολλές, ε, όπως είναι η γεωργική πολιτική. Έχουμε το πρασίνισμα, έχουμε τα ανώτατα όρια, έχουμε την σύγκληση των πληρωμών, αλλά αυτό δεν σημαίνει θεμελιώδη αλλαγή της πολιτικής. Και επίσης τα νούμερα πάνω κάτω διατηρούνται. Υπάρχει μια σχετικά, σχετική μείωση του μεριδίου της γεωργικής πολιτικής σε σχέση με το γενικό προπολογισμό, αλλά σε σύγκριση με άλλες πολιτικές η γεωργική είναι πολύ σταθερή, πολύ πιο σταθερή. Αυτά που βλέπουμε στην πρόταση λοιπόν της Κομισιόν σημαίνει πως δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για την πολιτική. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και εδώ η δική σας επιτροπή πρέπει να το συζητήσει. Δεν είμαστε εμείς ε, αρμόδιοι για να ε, μιλήσουμε για την ίδια την πολιτική. Πρέπει αυτό το ζήτημα να αναφερθεί και στο Συμβούλιο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για νούμερα. Πρέπει να συζητήσουμε για πολιτικές και αυτό το λέμε σε κάθε συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την Προεδρία. Για τα ποσά. Έχουμε κάποια σχετικά ποσά. Έχουμε την έκθεση ΣΟΥΡ όπου λέμε ότι δεν συμφωνούμε στην μείωση των κονδυλίων σε σύγκριση με το πολιτέ πλαισιο πλαίσιο 2007-2013. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν για τα ποσά. Έχουμε πάνω κάτω μια ιδέα. Όμως υπάρχουν πράγματα που δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα. Ο κύριος Κότα ανέφερε τον αποπληθωριστή. Αυτό δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί. Είναι κάτι το οποίο θα είναι μια θεσμική συμφωνία που θα την διαπραγματευτούμε είναι τμήμα του πακέτου του πολιετού πλαισίου, αλλά τα κάτι μελη ήδη δίνουν μηνύματα ότι δεν πρόκειται εύκολα να συμφωνήσουν με τον αποπληθωριστή, γιατί λένε ότι ο πληθωρισμός θα είναι λιγότερος. Χαμηλότερος. Αυτός ο αποπληθωριστής που είχαμε μέχρι στιγμής του 2% είναι ένα από τα θέματα που δεν είναι βέβαιο. Δεν έχει συμφωνηθεί. Έπειτα, Η ιδέα για το πώς το βάλουμε στην, όπως το βάλουμε στην έκθεση ΣΟΥΡ, ε, να έχουμε δηλαδή τις τιμές του 2013 συν τον αποπληθωριστή, αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Και στις συζητήσεις με το Συμβούλιο σε αυτή τη θέση επιμένουμε που έχει επισήμως ε, εγκριθεί εδώ. Αυτή είναι η βασική θέση του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και πάλι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο διαπραγματευτικό κοιτίον που θα έχουμε πιθανότατα τον Ιούνιο έτοιμο, που θα είναι τον Ιούνιο έτοιμο από το Συμβούλιο, θα έχουμε μια ιδέα ίσως χωρίς στοιχεία, ε, χωρίς νούμερα για τις πολιτικές. Αυτό που μας είπε το Συμβούλιο είναι ότι στο επόμενο Γενικό, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και μάλιστα η Ιδανική Προεδρία εντατικά εργάζεται για το πολίτες πλαίσιο θα ασχοληθούν με τα δύο μεγάλα ζητήματα, δηλαδή γεωργική πολιτική και πολιτική συνοχής και θα προσπαθήσουν να βρουν ε, συμφωνία για τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή οι προτεραιότητες, τρόπο χρηματοδότησης κτλ. χωρίς νούμερα και τον Απρίλιο-Μάιο θα συζητήσουν για τη γεωργία και για την συνοχή. Η κυρία Μαγκίνες ρώτησε το πού βρίσκεται το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο προσπαθεί να μην μένει απ' έξω Έχουμε το σύστημα της ενημέρωσης ε, πριν και μετά από το συνεδριάση του Συμβουλίου. Αύριο και μεθαύριο έχουμε συνεδρίαση με τη Δανική Προεδρία ακριβώς για αυτό το θέμα του πολιετούς πλαισίου. Έχουμε καλέσει εθνικούς βουλευτές, εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και ε, είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσουμε τις, δώσουμε μάλλον τις θέσεις μας. Και όπως σας είπα <coughs> υπάρχει και η δυνατότητα να μην συμφωνήσουμε. Αυτό θα σήμαινε, σύμφωνα με τα όσα είπε η Κομισιόν, ψηλότερο προπολογισμό. Αλλά πάλι εγώ δεν νομίζω, <coughs> γιατί το θέμα του τι θα γίνει μετά είναι πολύ κέριο, Νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Αν δεν κινηθεί το Συμβούλιο, έχουμε σαφώ πει και θα το ξαναπούμε αύριο και μεθαύριο και στα κρατημέλη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει διάθεσή του συν την απόρριψη του προπολογισμού. Αλλά και πάλι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη και υπάρχει μια ομάδα κρατών μελών που θέλει να μειώσει σαφώ περαιτέρω τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ότι θα πρέπει να συνδεθούν οι πολιτικές με τη χρηματοδότηση. Γιατί αν δούμε τον ευρωπαϊκό υπολογισμό τα τελευταία 20-30 χρόνια υπάρχει σχετική μείωση σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας και αύξηση των εθνικών προϋπολογισμών. Δηλαδή μετακινούμε τους πόρους από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο εθνικό. Ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Αυτό δεν είναι λογικό. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Για το χρονοδιάγραμμα ε, να πω ότι ιδανικά το πολιτές πλαίσιο θα πρέπει να συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του έτους αυτού, του τρέχοντος. Δηλαδή μετά από τη ιδανική προεδρία είναι η Κυπριακή. Πιθανότατα ο κύριος Φαρνορόμ Πόη θα παρέμβει στις διαπραγματεύσεις ως πρόεδρος του Συμβουλίου. Εγώ έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο θα κλείσουμε με τα τέλη του έτους, αλλά Όσο περισσότερο αναβάλλεται η τελική απόφαση, τόσο λιγότερος χρόνος θα υπάρξει στη διάθεσή μας για την ομαλή έναρξη του επομένου πολιτικού πλαισίου. Γιατί οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη πρέπει να προετοιμαθούν, να ετοιμάσουν κανονισμούς, νομοθεσίες κτλ. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να ξεκινήσει στις αρχές του 2014 η λειτουργία του νέου πολιτικού πλαισίου θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί νωρίτερα. Δεν τρέχουμε αυτά πάτε, θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά για την ώρα προτείνουμε ε, και στις συνομιλίες με το Συμβούλιο ε, ότι να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου τι μπορούμε να έχουμε συμφωνήσει. Βεβαίως, το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ πιο ισχυρό αν κρατήσουμε τις θέσεις μας και τις χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Να έχουμε τη συζήτηση δηλαδή για τις πολιτικές χωρίς τελική ψήφο, να έχουμε τη συζήτηση για τα νούμερα και έπειτα να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε με τον προπολογισμό ή αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθώσεις να μπορέσουμε να τις κάνουμε. Πραγματικά λοιπόν εκτιμούμε το την συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο, ώστε να μην αρχίσουμε να ψηφίζουμε χωριστές συμφωνίες στην Ολομέλη, γιατί κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει την θέση μας. Για την ευελιξία, Ο κύριος Δαντά είπε κάτι πολύ σημαντικό για τη δυνατότητα νέου χρήσης των κονδυλίων. Πολύ ευχαρίστως το, το θέλαμε. Η ευελιξία είναι ένα από τα θέματα που θέσαμε στο Συμβούλιο και το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό. Το Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι πολύ ενθουσιώδης για την χρήση της ευελιξίας και τον, για το να επιτρέψει τη νέα χρήση των κονδυλίων που δεν έχουν δαπανηθεί στον προπολογισμό. Αλλά είναι μια από τις θέσεις που θέλουμε να υπερασπιστούμε. Αν έχεις λιγότερα χρήματα και λιγότερα κονδύλια, πρέπει να είσαι πιο ευέλικτος για να μπορείς να προσαρμοστείς ε, και να πετύχεις τις πολιτικές σου. Και μάλιστα αυτό είναι κάτι που μπορείτε να προτείνετε άμεσα για τη γεωργική πολιτική, για το πώς δηλαδή θα εξασφαλιστεί αυτή η ευελιξία. Αλλά ως θέμα αρχής θα πρέπει να επιμείνουμε στην ευελιξία μέσα στην διαπραγματευτική ομάδα. Και κάποια ερωτήματα που θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Για τα ερωτήματα του κυρίου ε, του, Γιάρ, την το σύστημα της εξαίρεσης, η Κομισιόν προτείνει να καταργηθεί και να κινηθούμε σε ένα άλλο σύστημα κατά ποσών στα κρατημέλη. Αυτό θα είναι καυτό θέμα στο Συμβούλιο, όχι στο Κοινοβούλιο, γιατί στο Κοινοβούλιο είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά αυτό το περίπλοκο σύστημα των εξαιρέσεων και γι' αυτό επιμένουμε για τους ίδιους σπόρους και για ένα πολύ πιο διαφανές και ξεκάθαρο σύστημα για την χρηματοδότηση του προπολογισμού, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το Συμβούλιο, θα αποφασίσει εκείνο. Για τον αποπληθωριστή το ανέφερα. το θέμα για τις εθνικές, εθνικούς διοικητικούς μηχανισμούς, αυτό σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους εθνικούς διοικητικούς μηχανισμούς, αλλά αν αργήσουμε πολύ θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι εθνικές ε, ε, αρχές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά γρήγορες ε, όπως και οι ευρωπαϊκές αρχές για να ξεκινήσει καλά το πολιετές πλαίσιο. Δεν ξεκίνησε καλά το τρέχον γιατί πολλοί κανονισμοί ήρθαν αργότερα και γι' αυτό και αν δείτε την ε, απελευθέρωση των κοδηλίων στις αρχές του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου υπήρξε μεγάλη μείωση και αυτό δεν χρειάζεται το 2014 να ξαναγίνει γιατί θα χρειαστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να βοηθηθεί η έξοδος από την κρίση. Αυτά δεν ξέρω αν ο κύριος Μπέγκε θέλει να συμπληρώσει. Εγώ αυτά είχα να πω. Παρακαλώ, Ράιμερ. Ναι, συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Καλφίν. Όντως, η κατάσταση, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να μείνει, είναι ότι το κοινοβούλιο είναι ισχυρό όταν μπορεί στην πραγματεύση να μιλάει με μία φωνή. Και στην έκθεση σου. Είχαμε ευρύτατη συμφωνία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Στο Συμβούλιο έχουμε τους φίλους της συνοχής, τους φίλους της γεωργικής πολιτικής και τους φίλους της σφιχτής τσέπης. Και άρα και πολλούς άλλους μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε θέση πιστεύω ως Κοινοβούλιο να τοποθετηθούμε, να πούμε ποιες είναι οι θέσεις μας, να διαπραγματευτούμε αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα τα χρονικά. Και γιατί δεν θέλω να επαναληφθεί, όπως έχει συμβεί άλλη φορά, να αποφασίσει στη δεύτερη φάση του Συμβούλου ομόφωνα και τη στιγμή που αποφασίσει το Συμβούλιο η Επιτροπή με την πλειοψηφία να μην έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να πιέσει το Κοινοβούλιο για να λάβει μια απόφαση και να εξοικονομήσει έτσι χρόνο, χωρίς όμως κανένα περιθώριο για διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το σημείο το οποίο θέλω εδώ να αναφέρω ξεκάθαρα ενώπιον σα, ενώπιον τη Επιτροπή σα, ότι από την Επιτροπή αναμένω ξεκάθαρα μηνύματα, σαφή μηνύματα, πολύ σαφίστερα από ό,τι στο παρελθόν, ότι είναι διατεθειμένοι προτεραιότητε τι οποίε η ίδια έχει ορίσει και στι πληρωμέ και στο περιεχόμενο των μέτρων να τα στηρίξει, να τα διεκδικήσει και αν υπάρξει αντιπαράθεση να είναι στο πλευρό του Κοινοβουλίου και όχι να ε, υποχωρήσει ενώπιον του Συμβουλίου. Top down, bottom up. Η Πολωνική Προεδρία είχε προτιμήσει την προσέγγιση bottom up, η Δανική το top down ίσως θέλει με τον τρόπο αυτόν να ε, υποχρεώσει τα κράτη-μέλη σε κάποια αντίδραση. Εν πάση περιπτώσει, η συνοχή, η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, η γεωργία είναι σοβαρά ε, κεφάλαια στην πολιτική μας, κεφάλαια στα οποία έχουμε κοινέ δράσεις, έχουμε συναπόφαση και έχουμε να διαμορφώσουμε από κοινού τα μέτρα. Από την άλλη, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να συζητούμε για περιεχόμενο και δράσεις όταν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε προσέγγιση ως προς τα ποσά τα οποία θα διατεθούν. Και άρα υπό κάποιες, θα έλεγα, επιφυλάξεις μπορούμε να συστήσουμε ή μη τι άλλο προτεραιότητες, κάποια γενικά κεφάλαια. Όπως είχαμε πει και στη Σούρε, 12 συν, 2, συν 5 συν 2. Και να ορίσουμε και αρνητικέ προτεραιότητε. Αυτό παρακαλώ και σα ορίστε τι αρνητικέ προτεραιότητε βάσει των οποίων θα προσδορίσουμε την ημερήσια διάταξη. Ε, το πρόγραμμα δηλαδή που θα προβάλλουμε στο Συμβούλιο έρευνα, τεχνολογία, 30 δις λείπουν από την Ευρώπη για την, ε, για την Αζέντα 2020 τεχνολογία και την έρευνα. 0,7% στην αναπτυξιακή πολιτική που μόνο λίγα κράτη-μέλη υπηρετούν, ε, ικανοποιούν τις δεσμεύσεις τους στην υπόθεση αυτή. Μας λείπουν 30 με 35 δισεκατομμύρια στο σύνολο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουμε. Πρέπει όμως να πούμε από την άλλη όταν έχουμε ένα προβλησμό ποιος θα τον ε, χρηματοδοτήσει, πώς θα γίνει η κατανομή και τι είδους προτεραιότητες θα έχουμε ορίσει. Και ανάλογα με τις προτεραιότητες αναλαμβάνουμε και την πολιτική ευθύνη, ρωτήσει φυσικά ταυτόχρονα ότι δεν είναι εύκολο για ε, κανένα θεσμικό όργανο να προσδιορίσει αρνητικές προτεραιότητες και μια και αύριο έχουμε και τους τουριστές από ό,τι ξέρω ε, θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα πιο συγκεκριμένα. Από την άλλη πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνομιλίες της με διάφορους υπουργούς έχει συζητήσει αλλά υποτιμώντας από ό,τι φαίνεται τις συνέπειες σε εθνικούς προπολογισμού, γιατί η κυρία Κάθριν Τέιτ από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, φαίνεται να διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού της γεωργικής πολιτικής στη, στα προβλήματα της ε, γραφειοκρατίας. Και κάποιος υπουργός σήμερα μου είπε εμένα, και δεν ήταν γερμανός υπουργός, ε, πρέπει να σας επισημάνω, ότι για τη γεωργική πολιτική υπολογίζει από την εξοικονόμηση της, ε, σε γραφειοκρατία να κερδίσει, να εξοικονομήσει 50%, το 50% του προπολογισμού. Εν πάση περιπτώσει όμως, να σας πω τι γίνεται όταν έχετε μια προεδρία που θα ακολουθεί την ε, πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει το καθήκον βεβαίω η Προεδρία να ε, κάνει μια προσπάθεια να, να ξεύρει λύσεις, να προωθήσει αποφάσεις κτλ. Ωστόσο, πρέπει πάνω απ' όλα να μεριμνήσουμε έτσι ώστε ε, χειρισμοί σε επίπεδο συμβουλίου να μην θέσουν εκτός ε, εφαρμογής, να μην εξεδετερώσουν δηλαδή την εφαρμογή του Συμβουλίου του, της Συνθήκης της Λισαβόνας και γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε να είναι στο πλευρό του Κοινοβουλίου. Ενώ στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία μπορεί να λένε ότι θα ήθελα να συμμετέχει πιο εντατικά το, το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις, ενώ κάποια, άλλη, κάποια άλλα δεν επιθυμούν καθόλου συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Φαίνεται ότι ούτε από το Άκτο, ούτε από το ΣΟΥΙΦΤ, ούτε από το Μαρόκο μάθανε τίποτα ότι τα κράτη αυτά, δηλαδή δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι το Κοινοβούλιο έχει με σοβαρότητα πάντα αντιμετωπίσει τις ευθύνες του κυρίως σε περίπτωση συναπόφασης. Αυτό λοιπόν καλό τους διάφορου πολιτικού να το αντιληφθούν και ε, είναι καλό να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση ή αν το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι μπορεί με τη διαδικασία της συμφωνή νόμης, γιατί μόνο ναι ή όχι μπορούμε να πούμε χωρί τροπολογίε, δηλαδή να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το κείμενο, ε, μόνο ε, να δει αν θέλει να περιοριστεί σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, Πολιτικό συμβασμό είναι ότι λέμε 2013 στην, Ευρωπα... στην πολιτική με απόλυτους όρους, σε απόλυτους όρους διατηρούνται τα, ποσά, τα Αυτό έχουμε πει. Αυτό θέλουμε, θέλουμε τα ποσά 2007-2013 τη γεωργική πολιτική και αυτό είναι το μέγιστο σε πολιτικό συμβασμό που μπορούμε να δεχθούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άλλες αλλαγές ή εξελίξεις. Θα προτιμούσα όμως να μην ανοίξει αυτό το βαρέλι χωρίς πάτο. Διότι πια θα έχουμε χάσει κάθε δυνατότητα για να προσδιορίσουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία των μέτρων. Επίσης θα συμφωνήσω με τον κύριο Τέν για το outsourcing και για τα συγκεκριμένα προγράμματα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και παγκοσμιοποιημένε ε, συνέπειε για την γεωργική πολιτική την παγκόσμια οικονομία, είναι νομίζω λύσεις όπως το outsourcing που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίοι ουσιαστικά παραβιάζουν και τις αρχές της, της πολιτική ε, πολιτικής και αμφισβητούν την ε, χρηματοδότηση μέσω της κοινοτικής μεθόδου, μεθόδου 15, 17, 20 κράτη-μέλη, όσο και να είναι, πάντοτε είναι επικίνδυνο να μπούμε σε αυτήν την ατραπό. Και κλείνοντα, κύριε Πρόεδρε για το χρονοδιάγραμμα, οι προγνώσει μου φαίνονται πολύ δύσκολε. Πάντως να τα καταφέρουμε, αν δεν μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε αποφασιστική πρόοδο από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο και ω προ τα ποσά, αλλά και για την προκαταρκτική διαπραγμάτευση, προκαταρκτική συζήτηση για το περιεχόμενο, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αλλά, αλλά, λέω και προκαταλαμβάνω ίσως, ότι αν δεν υπάρξει άλλη λύση από, την, ε, από το 2013, από τα ποσά του 2013, κυρίε και κύριοι, ας μείνουμε στα ποσά του 2013. Μπορούμε. Απλώς πρέπει να ρυθμίσουμε τις νομικές βάσεις, αλλιώς κρίση τεράστια δεν, δεν θα προκύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εν πάση περιπτώσει Δεν υπάρχει λόγος να παρασυρώμαστε ή να αφήνουμε να μας οδηγούν σε αντιδράσεις ε, πανικόβλητες ορισμένοι από το Συμβούλιο από την Επιτροπή. Κανένας λόγος. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτά θα περιοριστώ. Τους επόμενους, τις επόμενες εβδομάδες μήνες θα συζητήσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Θα διατηρήσουμε βεβαίω τις ε, σχέσεις μαζί σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και για τα ποσά και για τα περιεχόμενα εδώ στο βαθμό που είναι δυνατόν να καταστήσουμε σαφές ε, το ποια είναι η θέση μας, δε για το Συμβούλιο. Νομίζω ότι ε, θα ληφθεί, ελπίζω ότι θα ληφθεί υπόψη με σοβαρότητα η θέση του Κοινοβουλίου και παρακαλώ το Συμβούλιο να αναλογιστεί με σοβαρότητα τη συνέπεια της όποιας επιλογής του. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε και τη Σοφία των συναδέρφων από τον προπολογισμό και βλέπουμε ότι πολλά από τα επιχείρηματά τους είναι κοντά στα δικά μας. Οπότε ελπίζουμε, παρόλο που θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, ότι θα πετύχουμε γιατί έχουμε μια γερή διαπραγματευτική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τον κύριο Κάλφεν και τον κύριο Πόκε για την συμμετοχή τους εδώ. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλος το λόγο. Ε, οπότε Κλείνει το σημείο αυτό, έχοντας ευχαριστήσει και τον κύριο Σκοντά και τον κύριο Λόγκο. Τώρα, περνάμε στο επόμενο σημείο στην εμμυρίσια διάταξη, που είναι το σημείο του Λουίς Μανουέλ Κάπουλα Σάντος, Α, όχι ακόμα αυτό. Έχουμε την παρουσίαση της μελέτης για την ελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελοϊνικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον καθηγητή Φεντάριση και την κυρία Φερντόνε. τον Αντώνιο Πέσερ, και τον κύριο Ντελάκουελ και τον Βιτσίσο Σεκουίνο από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονομίας από την Ιταλία. Είκοσι λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να παρουσιάσετε την μελέτη σας και μετά θα συζητήσουμε, θα κάνουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι κλπ. Λοιπόν, η κύριε Φερντόνε πρώτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Πολύ χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής της ΙΝΑ από κοινού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μοπελιέ της Πάδοβας και με τη συνεργασία επιπλέον υπερογνωμόνων του τομέα. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε στα πλαίσια μιας γενικότερης ανάλυσης για την οργάνωση, την κατάσταση του αμπελοινικου τομέα. Η αγορά του τομέα αυτού έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια και έχουμε περάσει από δομές που ήταν καθαρά γεωργικές σε μία δομή που διακόπτει η ομιλήτρια σε μία αγορά λοιπόν πιο διαρθρωμένη και που έχει να κάνει περισσότερο με την παραγωγή τροφίμων. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η αγορά του ίνου χαρακτηρίζεται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε ειδικού τομείς της αγοράς και που εξελίσσονται εντελώ διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν πρέπει όμως από την άλλη μεριά να πέσουμε στη βαγίδα και να νομίζουμε ότι δεν έχουν και καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί ακόμα και αν υπάρχει κατακαιρματισμό στην αγορά, παρόλα αυτά υπάρχει σύνδεση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Η κατανάλωση ίνου αυξήθηκε στις παραδοσιακά μη παραγωγές χώρες και μειώθηκε στις χώρες που παραδοσιακά παρήγαν ίνο. Η εμπορία έχει αυξηθεί και υπάρχει μια αύξηση ιδιαίτερα ψηλή, κυρίως στις ε, χώρες που πρόσφατα παράγουν ίνο. Υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή σκηνή. Βλέπουμε ότι οι νέοι παραγωγοί έχουν μεγάλη προσφορά, ενώ ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, έχουν ε, εξαίρετες επιδόσεις. Παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, ο πελοϊνικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαφέρει πολύ από τους νέους παραγωγούς όσον αφορά τη στρατηγική που ακολουθούν ή τη δομή μέσα στην οποία δουλεύουν. Και αυτό γιατί και στις δύο περιοχές υπάρχουν πάρα πολλές μικρές ε, και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και μάλλον λίγες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που είναι εξωπρόσεκτο επίσης είναι ότι υπάρχουν πολλές πολυεθνικές του τομέα που έχουν ε, μονάδες παραγωγής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις νέες ε, παραγωγούς χώρες. Έχοντα αναλύσει λοιπόν τη δομή της αγοράς, η μελέτη αυτή ανέλησε και τους μηχανισμούς λειτουργίας του συστήματος όσον αφορά τα δικαιώματα φύτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι ε, μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ότι υπάρχει διαφορετική προσαρμογή στις διάφορες χώρες, ανάλογα με τη σημασία και τον δυναμισμό που έχει ο αμπελοϊνικός τομέας στην ε, κάθε περιοχή που εξετάσαμε. Το σύστημα φύτευσης δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητά του ανάλογα με τα κράτη, τις περιοχές όπου αυτό αναλύθηκε. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο μηχανισμός μεταφοράς του δικαιώματος φύτευσης, γιατί οι διάφορες χώρες ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου εκ των προτέρων χρειάζεται αδειοδότηση ή υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης ελευθερία κυκλοφορίας. Ενώ αλλού υπάρχουν ποσοστώσεις για τον όγκο ε, ανταλλαγών μεταξύ ε, διαφορετικών ζωνών ή διαφορετικών τύπων ίνου. Διαφορές λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στην αγορά αλλά υπάρχουν και στις τιμές. Αναλύσαμε και εδώ την κατάσταση με ερωτηματολόγιο το οποίο στείλαμε σε διαφορούς φορείς και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την τιμή του δικαιώματος φύτευσης. Μάλιστα, η διαχείριση ε, γίνεται μερικές φορές από την ελεύθερη αγορά, αλλά τελικά και οι εθνικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει τις τιμές αυτές καθ' Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα διαπιστώσαμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο και το κόστος ε, του ενδιάμεσου που και αυτό με τη σειρά του διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το πώς γίνεται η διαχείριση του κόστους αυτού. Φαίνεται ότι το σύστημα δικαιώματος ε, φύτευσης δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην επέκταση των πιο δυναμικών επιχειρήσεων που θέλησαν να μεγαλώσουν την παραγωγή τους. Όμως η αγορά ε, Δικαιώματο φύτευσης δεν έχει μεγάλη διαφάνεια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στα κράτη-μέλη ή σε περιφέρειες όπου δεν είναι γνωστό ποιοι είναι εκείνοι που πουλούν ή που αγοράζουν ή που μεταφέρουν τα δικαιώματα αυτά φύτευση ή και προ όφελο ποιας επιφάνειας γίνεται αυτό. Ένα άλλο, κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει σαφέ είναι ότι υπάρχει κερδοσκοπία στις τιμές δικαιωμάτων κάτω από ορισμένες συνθήκες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για ένα σημαντικό εμπόδιο στην επέκταση της αγοράς. Η μελέτη μας προσπάθησε επίσης να κάνει μια εκτίμηση του σχήματος των φυτεύσεων με βάση την εξέλιξη των επιφανειών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εσωτερικό των βασικών ανταγωνιστικών χωρών της Ένωσης. Έτσι ανατρέξαμε σε ένα συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τον, τις επιφάνειες που έχουν φυτευθεί από κλίματα και τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά και που αντιπροσωπεύονται από τις τιμές ε, των εξαγωγών. Το συγκριτικό αποτέλεσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, φυτεύσεις στον νέο κόσμο, σίγουρα για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένωσης οι τιμές ε, συμπεριλαμβάνουν τις επιπλέον επιφάνειες που καλλιεργούνται ε, με κλίματα. Αν και πολύ συχνά υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, μια διαφορά ανάμεσα στην πραγματική φύτευση και την ε, πραγματική φύτευση και καλλιέργεια αυτών των κλιμάτων. Βρισκόμαστε σε ένα σύστημα συγκεκριμένων ποσοστοποιημένων δικαιωμάτων, γιατί πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει πλήρως να χρησιμοποιήσει το δυναμικό παραγωγής της οι επιπτώσεις των τιμών στις εξαγωγές στο, σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να παίζει λιγότερο σημαντικό ρόλο κυρίως για την ε, υπερπαραγωγή που έχει χαρακτηρίσει το παραγωγικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών καθώς και την επίπτωση ενός υψηλού επίπεδου εσωτερικής κατανάλωσης σε σχέση με την συνολική παραγωγή. Ωστόσο, συνολικά το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε αποδεικνύει ότι στις χώρες εκτός Ένωση η διάσταση της προσφοράς είναι σίγουρα πιο στενά συνδεδεμένη με την αγορά και στήνει να προσαρμόζεται, αν και με κάποια καθυστέρηση, στην ε, ε, προσφορά που υπάρχει από την ίδια την αγορά. Ε, ο αντίκτυπο των δικαιωμάτων φύτευση έχει εκτιμηθεί και με βάση μια συγκριτική μελέτη που έχει κάνει η βάση, η βάση δεδομένων της ε, ε, FADN. Αυτή δείχνει ότι η παραγωγή κρασιού με βάση τα κλίματα που έχουν ε, φυτευθεί δείχνει μεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης από ό,τι άλλες καλλιέργειες. Σχεδόν σε όλες τις ε, περιοχές που αναλύθηκαν μέσα στο πλαίσιο αυτής της μελέτης και αυτό κατά κάποιο τρόπο μας υποδεικνύει ότι μπορεί σε περίπτωση απελευθέρωσης να υπάρξει μια λανθάνουσα πίεση προς ε, μια αύξηση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ε, στα φιλιών. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των τιμών, τις εξελίξεις στις τιμές που θα έχουν υπάρξει εντωμεταξύ Ένα άλλο μαθηματικό μοντέλο προγραμματισμού και θετικής ε, θετικού μαθηματικού προγραμματισμού έχει οδηγήσει στην εκτίμηση αυτής της πίεσης αν και θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτό το μοντέλο και τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά δεν, καταφέρουν, δεν καταφέρνει να λάβει υπόψη καταλήλως τον κίνδυνο τον επενδυτικό και τις ε, χρηματοπιστωτικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με την ετήσια καλλιέργεια. Εν πάση περιπτώσει η FADN δείχνει πως η κερδοφορία υπάρχει και αυτό μπορεί να οδηγήσει προς νέα, ε, νέες καλλιέργειες κλιμάτων. Έπειτα η μελέτη στάθηκε στην εξέλιξη των πολιτικών που σχετίζονται με τις ε, φυτεύσεις για χώρες που δεν λειτουργούν με συνθήκες παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλο μέρος αυτών των χωρών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ίσω να υπήρξε παλιότερα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές περιορισμού και μάλιστα ορισμένες από αυτές τις χώρες τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σημαντικές κρίσεις υπερπαραγωγής. Στη συνέχεια, πριν προβεί στην ανάλυση των δύο επιλογών μεταρρύθμισης που είχαμε να μελετήσουμε, ξεκινάμε την αρχική ανάλυση της κατάστασης της εφαρμογής της ΚΟΑ του κρασιού που εγκρίθηκε το 2008. Η ανάλυση αυτών των πρώτων ετών εφαρμογής τονίζει τη δυσκολία εφαρμογής κάποιων ειδικών νέων μέτρων με ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα των αμοιβαίων ταμείων, τις ασφαλίσεις ε, για την ε, συγκομιδή και τα μέτρα της πράσινης συγκομιδής. Επίσης ε, τονίζει τη σημαντική την σημασία των παλαιών μέτρων που βρίσκονται στο phasing out και που θα ολοκληρωθεί η χρήση τους μέσα στο 2012 και μέσα στο πλαίσιο της ΚΟΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, την απόσταξη. Ε, επίσης ε, αναγνωρίζεται πως ε, στον συγκεκριμένο τομέα δεν παίζει μεγάλο ρόλο, ε, τόσο μεγάλο, το σχήμα της ενιαίας ε, ε, της μοναδικής μάλλον πληρωμής, της άμεσης πληρωμής που έχει επηρεάσει πολύ τους υπόλοιπους αγροτικής τομείς. Ενώ στο πλαίσιο της ΚΟΑ αυτός ο προγραμματισμός καλύπτει τη συνολική περίοδο την δημοσιονομική. Τώρα, ας μπούμε στην ουσία της πρώτης επιλογής που εμείς αναλύσαμε, που είναι αυτή που μιλάει για τις πιθανές επιπτώσεις ε, της ε, προτινόμενης κατάργησης των δικαιωμάτων φύτευσης προκύπτει ότι αν επιβεβαιωθεί αυτή η απόφαση για κατάργηση μετά το 2015 αυτού του μηχανισμού ελέγχου των επιφανειών, το μεγαλύτερο τμήμα των μέτρων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης για τον αμπελοϊνικό τομέα μπορούν άμεσα ή έμεσα να είναι χρήσιμοι στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα έχει στόχο την διακυβέρνηση του τομέα μετά από την κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πολύ σημαντικό, σημαντική η αξιολόγηση της ε, επιρροής ορισμένων αυτών των μέτρων παρέμβασης ε, και κυρίως των πιο πρόσφατων. Και μέσα στη μελέτη παρουσιάζονται και προτείνονται κάποιες ε, ε, προτάσεις για μια μεταρρύθμιση για μια αναθεώρηση όσον αφορά την προώθηση, τις επενδύσεις ε, και τις ασφαλίσεις ε, όσον αφορά την ε, συγκομιδή. Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις που είναι επιτάπητος για την ενιαία ΚΟΑ στην ουσία επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά για τον αμπιλενικό τομέα τους μηχανισμούς πληρωμών που υπάρχουν ήδη χωρίς να εξασφαλίζεται οποιοδήποτε συντονισμός με τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς στο πλαίσιο των ε, μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπάρχει βέβαια ο λανθάνων κίνδυνος ε, υπερπαραγωγής που συνδέεται με την κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξη, αλλά και στο πλαίσιο της ε, ΚΟΑ ίνου να, θα πρέπει να εισαχθούν και μέτρα ρυθμιστικά όπως όσον αφορά τον εμπλουτισμό, όπως όσον αφορά τι ενώσει παραγωγών και τι ε, κλαδικέ οργανώσει, γιατί θα χρειαστεί να ενισχυθούν ε, σημαντικά σε σχέση με τον ισχύοντα μηχανισμό, ώστε να ασκήσουν ένα ρόλο παρόμοιο με αυτόν που έχουν, για παράδειγμα, στον τομέα των οποροκυπευτικών. Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση μιας απελευθέρωσης, για να μπορέσουμε να έχουμε και να παρακολουθήσουμε τη δυνατή ε, εξέλιξη της παραγωγής θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα παρακολούθησης της φύτευσης των νέων κλιμάτων, γιατί έτσι θα μπορούμε να έχουμε ένα σίγουρο σύστημα για την ευρωπαϊκή παραγωγή, επί τη βάση του οποίου να ε, προβούμε σε διαδοχικές εκτιμήσεις. Ε, εδώ στην πυραμίδα αυτή βλέπετε στην ουσία την ε, λειτουργία της ΚΟΑ και είναι εύκολο έτσι να καταλάβουμε τι θα μείνει από αυτή την ΚΟΑ, γιατί θα έχουμε ένα σύνολο μέτρων phasing out που θα πρέπει να εξαφανιστεί, εξαφανιστούν μετά το 2015 το σύστημα ελέγχου δυναμικού, δηλαδή το καθεστώς αυτό ήδη καταργηθήκε φέτος και έτσι θα έχουμε ε, αυτά τα μέτρα που βλέπετε τώρα για την ΚΟΑΛΑ. Για να μπορέσουν να ισχύσουν αυτά τα μέτρα θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στα αριθμιστικά μέτρα, δηλαδή στους κανόνες ετικετοθεσίας, στο ρόλο ε, των ενώσεων των παραγωγών και αν αυτά τα μέτρα δεν ενημερωθούν η μελλοντική ΚΟΑ θα χρειαστεί να λειτουργήσει με μια αντίστροφη πυραμίδα όπου τα βασικά μέτρα δεν θα έχουν ε, κάποιες, ε, ε, δεν θα έχουν κονδύλια και δεν θα μπορούν να χειριστούν τον αντίκτυπο της διαδικασίας απελευθέρωσης. Και άρα θα είναι απαραίτητο να αντιστραφεί η πυραμίδα. Αντίθετα στην περίπτωση της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης, Σίγουρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από δύο σκέψεις. Η μία είναι η δυνατότητα επανεξέτασης της ε, απόφασης για την ε, κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης. Πρώτον, γιατί αυτό το μέτρο είχε τη δυνατότητα να συμβάλλει στον έλεγχο της παραγωγής χωρίς ε, να επιβαρύνει με κόστος τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και μάλιστα γεννώντας κάποιες θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τους καλλιεργητές που αποφασίζουν να σταματήσουν την παραγωγή έπειτα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από το καθεστώ, το οποίο ε, συχνά συνοδεύεται από διατάξει είτε εθνικού τύπου είτε περιφερειακού τύπου, που στενά συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα, έχει, έχουν τονίσει ε, ενάρετους μηχανισμούς μηχανισμού οι οποίοι ε, οδήγησαν σε επιτυχία και θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση έμπνευση για την αναθεώρηση της λειτουργία τη συγκεκριμένη ΚΟΑ. Σίγουρα η διατήρηση αυτού του σχήματος θα πρέπει να βασιστεί σε μια υπόθεση αναθεώρησή του όσον αφορά τη λειτουργία του, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις πιο σημαντικές, ε, τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα και δυσλειτουργίε και για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του δυναμικού παραγωγή. Η δομή του νέου συστήματο θα πρέπει να βασιστεί σε δύο πυλώνες. Ένα θα είναι η βελτιωμένη αγορά όσον αφορά του κανόνε λειτουργία και έναν, ε, μια περιοδική ε, αξιολόγηση που στόχο θα έχει να επανεξετάζει την ομαδοποιημένη διάσταση της παραγωγής ώστε να μπορέσει να επιτρέψει σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη ή περιοχές την αύξηση του δυναμικού τους. Αλλά για να βελτιωθεί ε, η αγορά των δικαιωμάτων φύτευσης είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν δύο πτυχές τουλάχιστον στις λειτουργίες τους. Οι τεχνικοί κανόνες για την ανταλλαγή των δικαιωμάτων φύτευσης και η δυνατότητα διεύρυνσης των ορίων αποδεκτών μεταφορών αυτών των δικαιωμάτων. Ναι, οι κανόνες στην αγορά θα ε, διευκόλυναν στην αποφυγή ε, κερδοσκοπίας, στο, αλλά και την αποφυγή του κινδύνου απατών. Επίσης θα μπορέσει να περιορίσει την, την υπερβολική διαφοροποίηση των τιμών που έχει περιορίσει τις μεταφορές σε συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά θα συμβάλλουν και στην μείωση του κόστους διαμεσολάβησης που ορισμένες φορές ήταν πολύ υψηλά. Εδώ η μελέτη στέκεται στην πρόταση εισαγωγής ενός συστήματος πληστηριασμών για την πώληση των δικαιωμάτων φύτευσης που εξάλλου είναι ένας μηχανισμός που έχει λειτουργήσει σε κάποιες χώρες. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της ε, ε, δημιουργίας μεγαλύτερων περιοχών ανταλλαγής για, και ενδεχομένως και ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο εντός του ιδίου κράτους. Η συζήτηση και τα έγγραφα στα οποία βρίσκει κανείς τις θέσεις που έχουν εκφραστεί, περισσότερο κλείνουν υπέρ τη διατήρησης του καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευση και στην αναθεώρησή του. Λιγότερε είναι οι θέσει υπέρ της κατάργησής του και της πλήρους απελευθέρωσης, αλλά... Η μελέτη αυτή δεν, έχει, δεν συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία, υποστηρίζοντα συγκεκριμένες ιδέε ή ε, ε κατευθύνσεις. Σίγουρα σχεδόν όλες αυτές οι μελέτες αναφέρονται σε μέτρα ελέγχου της παραγωγής, αλλά καμιά μελέτη δεν μπορεί να τα καθορίσει όλα αυτά με σαφήνεια. Πριν να φτάσουμε στα βασικά συμπεράσματα, πορίσματα σε σχέση με τις δύο επιλογές, που αναλύθηκαν, θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε ορισμένα θέματα κλειδιά που κατά τη γνώμη μας αποτελούν βασικά στοιχεία που θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του στην ανάλυση του θέματος αυτού. Καταρχήν, επειδή η ΚΟΑ είναι, ανέκαθεν είχε αναγνωριστεί ως μια ιδιαιτερότητα στο εσωτερικό της Κούγουπου, το θέμα των ε, δικαιωμάτων φύτευσης δεν θα πρέπει να κριθεί ως άτοπο σε ή άσχετο με τις κοινέ αρχές της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, ούτε ε, ότι οδηγεί σε συγκρούσεις σε σχέση με διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Μάλιστα, το πρόγραμμα δικαιωμάτων φύτευσης θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την πολιτική που σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ, με την πολιτική που αφορά την ονομασία προέλευσης, αλλά και ούτε και με άλλα, ε, προ, άλλους κανονισμούς που αφορούν τις κοινέ οργανώσεις αγορών. Όσον αφορά την πολιτική κατανάλωση υνοπνεύματων ποτών, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι σχεδόν σε όλε τι χώρε, τόσο τη Ένωση όσο και εκτό, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στι ε, δραστηριότητε διαφήμιση και πώληση του ίνου. Και άρα η υπόθεση απελευθέρωση θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να λάβει υπόψη τη συγκεκριμένη πτυχή. Και έπειτα είναι απαραίτητο και μάλιστα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας, να ξεχωρίσουμε δύο ερωτήματα τα οποία συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Το ένα είναι η γενική ρύθμιση των ε, δικαιωμάτων φύτευσης και το άλλο θέμα που αφορά τη ρύθμιση της ε, παραγωγής με ονομασία προέλευσης. Τα δύο αυτά θέματα μεταξύ τους διαφέρουν αν και δεν είναι απόλυτα ξεχωριστά, διότι είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η αγορά ίνου με ονομασία προέλευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί χωριστή τελείως αγορά από την υπόλοιπη αγορά των μπελονικών προϊόντων. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερόμαστε και σε αυτά τα προϊόντα, αλλά το θέμα των δικαιωμάτων φύτευσης δεν μπορεί αποκλειστικά να αφορά αυτή την κατηγορία ίνου και παραγωγής. Εν κατακλείδη, η μελέτη μας στόχο έχει να τονίσει ορισμένες πτυχές που σχετίζονται τόσο με την υπόθεση της απελευθέρωσης όσο και με αυτήν της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης. Όσον αφορά την απελευθέρωση είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς κάποια πλεονεκτήματα που μπορεί κανείς να αναμένει από μια τέτοια διαδικασία ε, ορισμένα όμως πράγματα συνδέονται με τους δυνητικούς κινδύνους και κατά πόσο αυτοί είναι δυνατόν να, να, αυτούς είναι δυνατόν να τους διαχειριστούμε και να περιορίσουμε αυτούς τους ε, υψηλούς κινδύνους. Κάθε μια από αυτές τις επιλογές φυσικά ε, φέρνει μαζί της διαφορετικούς προβληματισμούς όσον αφορά τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Σίγουρα με την απελευθέρωση, η απελευθέρωση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και μπορεί επίσης να επιτρέψει μια μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης από πλευράς της προσφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κρασιά με χαμηλότερες τιμές κυρίως. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα αυτά συνοδεύονται από έναν κίνδυνο απώλειας ελέγχου της, ε, του ελέγχου της παραγωγής, του δυναμικού της παραγωγής, εφόσον δεν, υπάρχει, δεν θα υπάρχει κατάλογος των αμπελονικών επιφανειών. Μπορούμε όμως αυτό να το διαχειριστούμε με την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης κινδύνου και με μέτρα αυτοελέγχου της παραγωγής τα οποία θα ασκήσουμε ασκούν οι ενώσεις παραγωγών. Ένας άλλος κίνδυνος είναι να σταλούν αντιφατικά μηνύματα στην αγορά και σε αυτό τον κίνδυνο μπορεί κανείς ε, να τον αναχαιτήσει εγγυόμενος τη σωστή παροχή ε, ορθών και ακριβών πληροφοριών για την παραγωγή που θα τίθεται στη διάθεση όλων των φορέων. Επίσης ε, υπάρχει ο κίνδυνος αποδυνάμωσης του ανταγωνιστικού ρόλου που έχουν κερδίσει διάφοροι φορείς του τομέα που δεν είναι αυτοί που λειτουργούν στα συγκεκριμένα προϊόντα αριστείας ή πολύ ειδικευμένα προϊόντα. Αυτό θα, μπορούσε να, θα μπορούσαμε να το αντιπαρέλθουμε εάν υπάρξουν ε, συγκεκριμένες μορφές ε, μέτρων για τον αμπελινικό τομέα και μέτρα για την διαχείριση της προσφοράς, τα οποία θα θέτουν σε εφαρμογή πάλι οι διεπαγγελματικές ε, οργανώσεις και ενώσεις. Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει η αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικονομικών ε, παραγόντων και απώλεια σταθερότητα σε απομακρυσμένες περιοχές. Και αυτά θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και από ένα ειδικό καθεστώς ε, ενιαίας πληρωμής. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο πλαίσιο της ε, ΚΟΑ Τώρα, αν αντιθέτως το, διατηρηθούν τα δικαιώματα φύτευσης, θα μπορούσε να προληφθεί υπερβολική προσφορά θα διατηρηθεί η δομή του αμπελονικού τομέα της Ευρώπης και μεγαλύτερη βιωσιμότητα για τις περιφερειακές και πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές. Εκεί βέβαια υπάρχουν και εκεί κίνδυνοι που συμπίπτουν ε, με την αποδυνάμωση της δυνατότητας αντίδρασης ε, του τομέα και σε αιτήματα που μπορεί να προέρχονται από την αγορά και εκεί θα μπορούσε ο τομέας να ανταποκριθεί με πιο ελαστική διαχείριση από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα για την χρήση του δυναμικού παραγωγής. Και σε αυτή την περίπτωση για να αποφυγεί, αποφευθεί μάλλον η λήψη αποφάσεων που δεν είναι βάσιμες θα μπορούσε να υπάρξει μια, ένα σωστό σύνολο πληροφοριών για την παραγωγή και για την πρόοδο και τις εξελίξεις στις αγορές. Αυτή την επιλογή βεβαίως θα μπορούσε να συνδεθεί και το θέμα μάλλον της αύξησης του κόστους παραγωγής όπου κανείς θα μπορούσε να το καταπολεμήσει μέσω της αγοράς ε, και των πληστηριασμών των δικαιωμάτων φύτευσης όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Επιπλέον αυτή η πολιτική θα ήταν πιο απλή στην εφαρμογή της από ότι η προηγούμενη, αλλά δεν πρέπει κανείς να υποτιμά την δυσκολία επίτευξης πολιτικής συμφωνίας σε σχέση με δυο συγκεκριμένες πτυχές, τις πιθανές αλλαγές στη διάσταση του δυναμικού παραγωγής και στον ορισμό της διάστασης των περιοχών ανταλλαγής των δικαιωμάτων φύτευσης. Στη διαδικασία ε, μεταφοράς των δικαιωμάτων φύτευσης. Εν κατακλείδη να σας πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η αγορά ίνου και ο τομέας του ίνου είναι τόσο περίπλοκη που είναι αδύνατον να φτάσει κανείς σε μια σαφώς εντοπισμένη βέλτιστη απόφαση που θα ακολουθεί τη δυνατότητα, τις δυνατότητες ε, και τη διατήρηση των ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών ίνου. Η απελευθέρωση βεβαίως θα μπορούσε να καταστήσει πιο δυναμική την προσφορά ίνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας χώρο κυρίως σε νέες επιλογές που συνδέονται με τις ενδείξεις της ποικιλία και των κλιμάτων και των ε, ε, χρονολογιών που θα υποδεικνύονται στις ετικέτες. Αν αυτή η αποφάση, απόφαση ληφθεί με, με ε, συνοδεία διάφορα αντισταθμιστικά μέτρα, δεν θα επιφέρει τραγικές ε, αλλαγές. Δεν θα έχει δηλαδή τραγικό αντίκτυπο για τον ε, μπελονικό τομέα στην Ευρώπη. Στόχος είναι να προστατευτεί καλύτερα η σημερινή δομή του αμπελονικού τομέα στην Ευρώπη, ε, προωθώντας ε, την παραδοσιακή μορφή προσφοράς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτή η επιλογή ακολουθηθεί από τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, δεν θα πρέπει να εμποδίσει την ανάπτυξη του αμπελονικού τομέα της Ευρώπης. Πολλά από τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία αποδεικνύονται σε σχέση με τη μία ή την άλλη επιλογή, θα πρέπει να εξεταστούν και να σταθμιστούν πολύ καλά, γιατί με βάση την επιλογή που θα γίνει μπορεί να οδηγήσουν στο σε μια βελτίωση των μέτρων στο πλαίσιο της ΚΟΑ για τον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, ε, ευκαιρία παίρνω εγώ εδώ να λαμβάνω την εξουσία μια που λείπει ο πρόεδρος. Ο κύριος Νταντά είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ κύριε Νταντά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια σε εκείνους που ετοίμασαν την ανάλυση αυτή, Πόντως εξετάζει όλες τις περιπτώσεις. Σπάνια λέμε μπράβο. Αλλά σε σχέση με τα διάφορα που έχουμε ακούσει για το θέμα, η δικιά σας δουλειά συνθέτει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε. Χθες το βράδυ, με πρωτοβουλία της κυρίας Λούλινγκ και μου του ιδίου, 350 άνθρωποι, ε, βρεθήκαμε να συζητήσουμε για αυτά ακριβώς τα θέματα. Υπήρχαν 8-9 υπουργοί, 30 βουλευτές από διάφορες χώρες για τα δικαιώματα φύτευσης, έτσι, από κάθε πολιτικό χρώμα. Ως εισηγητής, ε, λοιπόν, ε, εγώ ανέλαβα την χθεσινή οργάνωση εισηγητής για την σχετική ΚΟΑ. Νομίζω, λοιπόν, ότι το βασικό είναι ότι η ιδέα που προωθήθηκε είναι ότι πέρα από τις ε, μακροοικονομικές διαστάσεις, το θέμα της διαχείρισης του αμπελιού και της παραγωγής ίνου στην Ευρώπη, έτσι όπως τη γνωρίζουμε εδώ και 40 χρόνια, έχει έναν τριπλό στόχο που εγγράφεται στα πλαίσια της αεφόρου ανάπτυξης που θέλουμε σήμερα για την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα το αμπέλι παίζει και περιβαλλοντικό ρόλο, πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό ρόλο, γιατί ε, διαμορφώνει το τοπίο, γιατί αντιμετωπίζει την διάβρωση, αλλά έχει και μια κοινωνική διάσταση. Μια κοινωνική διάσταση, διπλή μάλιστα, και πολιτιστική, διότι το αμπέλι και το κρασί είναι μια πολιτιστική κληρονομιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη μεριά, με τον παραδοσιακό όρο κοινωνικό, έχει και άμεσες και έμεσες επιπτώσεις. Πολύ συχνά οι καλλιέργειες βρίσκονται σε πλαγιές και όχι στην πεδιάδα που είναι πιο εύκολη η διαχείριση εκεί. Κάποιος χτες είπε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο τελικά κατανέμει τον πλούτο ε, σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και είναι σωστό πιστεύω. Όντως, εδώ πέρα πρόκειται και για μια οικονομική διάσταση, διότι έχουμε τον τουρισμό. Όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργήσαμε την ιδιαιτερότητα των εδαφών μας. Τελικά πρόκειται για μια χωροτοξιακή διάσταση. Μπορέσαμε όμως να βελτιώσουμε και την ποιότητα των προϊόντων μας. Απόδειξη, ακόμα και οι τελευταίες χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που ακολουθούν 10 χρόνια περίπου τώρα την πολιτική αυτή, έχουν γίνει ποιοτικά άλματα. Η διαχείριση λοιπόν του συστήματος του αμπελιού αποτελεί και πηγή διαφοροποίησης. Και αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι αρνητική, αντίθετα είναι ένας τεράστιος πλούτος και για τον Ευρωπαίο καταναλωτή αλλά και για τις εξαγωγές μας. Και όταν λοιπόν η Ευρώπη αναρωτιέται ε, επειδή χάνει ε, και έχει λιγότερες εξαγωγές, με 20 δις ευρώ από τα μπέλια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η εξαγωγή αυτή και τι έσοδα μας προσφέρει. Πολύ σωστά υπογραμμίσατε ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε το σύστημα, δεν πρέπει να το διατηρήσουμε ακριβώς όσο έχει σήμερα. Γιατί τη διαχείριση των δικαιωμάτων φύτευσης, έτσι όπως εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες, καταλήγουν σε κανόνες κατά του ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να τα ξαναδούμε, πρέπει να επανορίσουμε τα δικαιώματα φύτευσης για να υπάρχει ένας πραγματικά ευρωπαϊκός κανόνας, ακόμα και αν η διαχείριση γίνεται αποκεντρωμένα. Τουλάχιστον εγώ προς αυτή την κατάφυνση σκοπεύω να δουλέψω ως εισηγητής για την κοινή οργάνωση αγοράς. Ευχαριστώ. The next speaker. Ευχαριστώ. Επόμενος είναι η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία όσον αφορά τα δικαιώματα φύτευση. Όντω, χθες το βράδυ είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνάντηση για τα δικαιώματα φύτευση και εγώ ήμουν εκεί εκ μέρου του ΕΛΚ. Αυτοί που λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε τα δικαιώματα αυτά φύτευση και ότι δεν χρειάζεται εξωτερική ρύθμιση για τον τομέα αυτό και ότι η αγορά από μόνη της θα μπορούσε να απορροφήσει ότι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο τομέας, δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Εγώ πιστεύω ότι τα δικαιώματα φύτευσης απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένα μέσο πολύ χρήσιμο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βοηθάει στο σχεδιασμό της παραγωγής με ένα οικονομικό και επιχειρηματικό σκέλος που έχει να κάνει με τις αμπελουινικές ε, επιχειρήσεις. Δεύτερον, απέδειξε ότι είναι πολύ χρήσιμος μηχανισμός για την πρόθεση της ποιότητας των ευρωπαϊκών κρασιών. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το πρασίνισμα, με τη διαχείριση των κινδύνων κλπ. κλπ. είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι ένα μέσο το οποίο απέδειξε και αυτούς τους δύο λόγους που σας εξήγησα πόσο χρήσιμο είναι. Και οικονομικά. Ορισμένοι λένε ότι η κερδοσκοπία στις τιμές μπορεί να έχει κάποια σχέση με αυτό. Με τα δικαιώματα δηλαδή φύτευσης και με την ανάπτυξη της αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι αντιφατικό ως προς διάφορες οικονομικές αναλύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί βλέπουμε ότι αυξάνει η εξαγωγή, αλλά έχουμε λιγότερες, ε, λιγότερο όγκο εμπορίας. Άρα δεν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι πρόκειται για κερδοσκοπία, πρόκειται για ρύθμιση της αγοράς. Επίσης, ορισμένοι λένε ότι υπάρχουν ε, θετικές επιπτώσεις από την ελευθέρωση σύντομα. Ούτε με αυτό συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις και μάλιστα αμέσως εφόσον ε, καταργηθούν τα δικαιώματα φύτευσης μέχρι το 2015 θα υπάρχουν επιπτώσεις και στο περιβάλλον, μεγάλες, σημαντικές και τραγικές. Γιατί ακριβώς στη, στα χειρότερα εδάφη φτιάχνουμε καλό κρασί. Και αν δεν φτιάχνουμε εκεί κρασί, να βάλουμε αμπέλια δηλαδή, τότε θα εγκαταλειφθούν τα εδάφη αυτά και θα υπάρξει απερίμωση που δεν τη θέλουμε δίνουμε χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Κορβανά για να αντιμετωπίσουμε την απερίμωση. Οπότε πρέπει να το ξανασκεφτούμε πριν πάρουμε ένα τέτοιο καταστροφικό περιβαλλοντικά μέτρο. Έπειτα θα υπάρξουν περισσότερα κοινωνικά προβλήματα ανεργίας και οικονομικής ύφεσης για πολλές ευρωπαϊκές περιοχές που δεν βρίσκομαστε βέβαια όπως καταλαβαίνετε και στην καλύτερη οικονομικά στιγμή τα δικαιώματα λοιπόν ε, φύτευσης πρέπει να ελέγχονται, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και να ελέγχονται και από τους παραγωγούς και από τη δημόσια δίκηση, όπως γίνεται και τώρα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την αϊφόρο ανάπτυξη. Το λένε οι επιχειρηματίες. Και πέτυχαν επίσης μια ισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά πολύ αποτελεσματική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υποστήριζε την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης. Τώρα λοιπόν ευτυχώς αλλάζει το Συμβούλιο Γεωργίας γιατί όλο και περισσότερες χώρες δείχνουν ότι θέλουν να διατηρηθούν τα δικαιώματα φύτευσης. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης είναι διατεθειμένη να το συζητήσει από τον Οκτώβριο ο επίτροπο Τσόρο μας το είπε στην Ολομέλεια. Οπότε αν προχωρήσουμε πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια συζήτηση καθαρά οικονομικής ελευθέρωσης, αλλά έχουμε να κάνουμε με την ε, χρήση των εδαφών, έχουμε να κάνουμε με ε, παραδόσεις και με την ύπεθρο, πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την γεωργική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόινινγκ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τους... Θέλω να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να πω ότι φαίνεται να προαγωνίζονται όλοι να διαφυλάξουν τη Γεωργία ενώ η Επιτροπή έχει πάρει να επιστρέψει τον δρόμο της φιλελευθεροποίησης, απελευθέρωσης. Όλοι λοιπόν προσπαθούν να διαφυλάξουν τα δικαιώματα φύτευση. Δεν είδα κανέναν ε, καλλιεργητή στη Γερμανία να λέει Α, πρέπει να μεριμνήσουμε για την απελευθέρωση τη αγορά. Άρα λοιπόν αυτοί που μιλούν ε, περί, περί διαφύλαξης ε, των μέτρων, περί διατήρησης των μέτρων, νομίζω ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Και Εάν προκύψει περισσότερη παραγωγή, ε, προφανώς οι πιέσεις στις αγορές θα έχουν σαν συνέπεια να έρθουν οι παραγωγοί εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται την πίεση πιο σκληρά να έρθουν σε εμά και να ζητήσουν επιδοτήσει, ενισχύσει, όπω άλλωστε έχουμε δει και στην περίπτωση του γάλακτο και σε άλλε περιπτώσει, με αποτέλεσμα τελικά να ε, αυξηθεί η επιβάρυνση για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Πρέπει επίση, εάν ε, ένα υπερουργό δεν μπορεί να παραγάγει ή, αν δεν μπορεί να καλλιεργήσει το αμπέλι του, θα πρέπει να του βρούμε και μια εναλλακτική. Ή διαφορετικά, εάν έχει πιο πολύ παραγωγή, θα πρέπει να βρούμε διέξοδο για τα προϊόντα του στην αγορά. Γιατί το αμπέλι δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από μια άλλη καλλιέργεια. Έτσι λοιπόν, η κατάσταση αλλάζει, το βλέπουμε, υπάρχουν κάποιε προθέσει ε, περί τροποποίηση των δεδομένων, αλλά νομίζω ότι ο σωστός δρόμος δεν είναι απελευθέρωση που προτείνει η Επιτροπή, αλλά μια πιο αυστηρή διαχείριση της αγοράς, μια πιο προστατευτική διαχείριση της αγοράς. Η ρύθμιση δηλαδή της αγοράς και έτσι ε, ουσιαστικά η δυνατότητα να προσφέρουμε στον ε, καλλιεργητή, στον αβελουργό ένα μέλλον στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κλάση. Βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει κανείς το βλέμμα του και να κοιτάξει το μέλλον. Με τις διάφορες παρατηρήσεις που ακούστηκαν βλέπουμε ότι θα είναι μάλλον ενδιαφέρον να ε, δούμε πού θα μας το οδηγήσουν όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι ορισμοί του εγγράφου μας δείχνουν ότι οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι, πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα διακυβεύονται εάν προχωρήσουμε στην, ε, ε, στις προτάσεις αυτές. Και ρωτώ για τα κονδύλια και την σχετική παρατήρηση, πώς καταλήγεται στο συμπερασμό όταν λέτε δηλαδή ότι η απελευθέρωση μπορεί να ε, ασκήσει πίεση για την αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας αμπελιού. Εγώ δεν ε, νομίζω ότι η προοπτική είναι η αύξηση των εκτάσεων, μάλλον είναι η μετατόπιση των εκτάσεων καμπελοκαλλιέργειας. Ο κύριος Χόισλινγκ γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι εξέθεσε πάρα πολύ καλά την ε, κατάσταση. διότι οι, οι πλαγιές πάνω στις οποίες καλλιεργείται το αμπέλι δεν προσφέρονται για άλλες ε, καλλιέργειες. Και έτσι τίθεται μεγάλο πρόβλημα αν μετατοπιστούν αυτές οι καλλιέργειες. Επίσης πολλά ερωτηματικά που μας απασχολούν ε, στη Γερμανία τουλάχιστον έχουν ήδη ρυθμιστεί ένα σαφές ε, καθεστώς το οποίο επιτρέπει στον αμπελουργό να κάνει τη δήλωσή του όταν αποφασίσει να κάνει νέα φύτευση. Ε, επίσης όταν προχωρεί σε εκρίζωση ή έχει ένα περιθώριο 8 ετών ε, που μπορεί να διατηρήσει το, την έκταση του, δηλαδή να διατηρήσει την, ε, στη διάθεση του την συγκεκριμένη έκταση, μετά την πάροδο των 8 ετών περνάει πάλι στο Εθνικό Μητρό ε, Βελονικό Μητρό. Επομένω, ε, είναι τα πράγματα πολύ καλά ρυθμισμένα στη Γερμανία και ρωτώ γιατί βλέπετε τέτοια δυσκολία προ τη ρύθμιση αντίστοιχα και στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικό δίκαιο. Διότι νομίζω ότι αν πρόκειται να κάνουμε κάποια τροποποίηση στην νομοθεσία ή μη τι άλλο, θα πρέπει να ελέγξουμε ότι δεν επιδεινώνονται οι συνθήκε σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία. Και πρέπει να πω ότι με ανησυχεί όταν λέτε ότι αποδεσμεύουμε τις εκτάσεις, μπορούμε να έχουμε περισσότερη παραγωγή και θα χρειαστούμε μέτρα αντικατάστασης. Ε, δηλαδή, επιστρέφουμε στα παλιά γνωστά εκείνα. Ε, μέτρα, τα οποία όμως εμείς τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία δεν έχουμε κανένα επιχείρημα για να τα υποστηρίξουμε. Γιατί ούτε ο καταναλωτής ούτε ο αμπελουργός θα δεχθούν αυτήν την ε, οπισθοδρόμηση προς τις παλές αγορές, τη ρύθμιση των αγορών, ε, τον έλεγχο στην απόσταξη και όλα αυτά. Πολλά λοιπόν θα γλιτώναμε εάν εγκαταλείπατε αυτή την πρόταση και όταν βλέπουμε μέτρα και μέτρα αντικατάσταση ε, των συνεπειών της, η αποκατάσταση των συνεπειών τη απελευθέρωση. μάλλον πρέπει να εισαγάγετε περισσότερα μέτρα για να αποκαταστήσετε τι ζημιές ε, τη απελευθέρωση παρά ε, αν αφήνατε τα πράγματα όπω έχουν τώρα. Λοιπόν, καλύτερα να τα αφήσουμε όπω είναι. Και ελπίζω να αντιληφθεί η Επιτροπή ότι είναι δύσκολα τα μέτρα που εισάγει. Συμφωνώ λοιπόν ω προ τα συμπεράσματά σα ότι πρέπει να διατηρηθούν τα δικαιώματα φύτευση. Ναι, πολλά είναι τα επιχειρήματα όμω τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον προβληματισμό αυτών για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων ε, φύτευσης. Η Επιτροπή, ο Επίτροπος δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνουν και να εισάγουν μέτρα παρά την αντίθετη βούληση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγγύηση και για την παραγωγή ίνου και για την επιβίωση όλων των περιφερειών αυτών. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο του τουρισμού μας, με ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καλό θα ήταν αυτό το μήνυμα να φτάσει μέχρι την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και που τόνισε ε, κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με το θέμα της διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης. Η συνάδελφος Κλάς ρώτησε χτες κατά πόσο υπάρχουν διαφορετικά, ε, διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης και φυσικά και υπάρχουν και εξαρτώνται κυρίως από την ευελιξία γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που περιορίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων από τη μια περιοχή στην άλλη ενώ σε άλλες χώρες αυτή η μεταφορά είναι σχετικά σχετικά εύκολη, δεν έχει και κανένα όριο. Αυτή είναι η βασική διαφορά και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να σκεφτούμε και εδώ, στο εσωτερικό της Επιτροπής μας, αυτό το στοιχείο. Γιατί όσο λιγότερο επιτρέπεται το να μεταφέρονται τα δικαιώματα από το ένα σημείο στο άλλο, τόσο περισσότερο το σύστημα προστατεύει ναι, μεν την ίδια την περιοχή, αλλά μετατρέπεται σε το σύστημα. Όσο πιο ευέλικτο είναι το σύστημα και επιτρέπει την μεταφορά από τη μια περιοχή στην άλλη, από τη μια περιφέρεια στην άλλη, ή και εσείς αναφέρατε και τη δυνατότητα μεταφορές από το ένα κράτος στο άλλο, τόσο περισσότερο ευέλικτο γίνεται το σύστημα και όπως είπατε η συνολική φυτευμένη ε, επιφάνεια μειώνεται ε, κάθε χρόνο. Ενώ αν το σύστημα ήταν πιο ευέλικτο, τόσο περισσότερο ίσως θα υπήρχαν και περισσότερες ε, φυτεύσεις. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή τι τελικά επιθυμούμε. Περισσότερη ευελιξία, είναι πιο σωστός ε, τρόπος, ε, πιο ευφύης τρόπος σε σχέση με την ε, άμεση εγκατάλειψη αυτού του συστήματος. Κάτι επίσης που είπατε σημαντικό είναι ότι η αγορά θα πρέπει να είναι διαφανής πιο διαφανής από ό,τι τώρα. Γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι σαφές, ότι εγώ υποστηρίζω και μιλώ για την Ιταλία το δικαίωμα φύτευσης ξεκινώντας από την Σικελία προς τη Βόρεια Ιταλία, το, η τιμή του τριπλασιάζεται. Και τα χρήματα αυτά δεν καταλήγουν στις τσέπες των καλλιεργητών, που εμπορε... αλλά στα στέπες αυτών που εμπορεύονται τα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μήπως θα μπορούσε να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα πληστηριασμών και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε ε, και θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο γιατί όσο γίνεται πιο ευέλικτο το σύστημα τόσο διαφανέστερη θα πρέπει να είναι και η αγορά. Γιατί όταν ένα δικαίωμα πάει από το ένα από τη μία καλλιέργεια στην άλλη, από το ένα σύστημα στο άλλο, ε, δεν διατηρείται πάντα εύκολα η διαφάνεια. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Thank you and, uh, Mrs. Ευχαριστούμε. Κυρία Λούλινγκ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι χθες... εξεπλάγην από Κάτι που είπε ο Γάλλος Υπουργό Γεωργίας, ο κύριος Ντοντάς, συνόψησε λίγο πολύ τι μας είπε σχετικά με την ε, καλή κατάσταση του αμπελοϊνικού τομέα. Αναρωτήθηκε όμως γιατί η Ευρώπη θέλει με μέτρα που δεν έχουμε σκεφτεί αρκετά, έτσι φαίνεται από τις διάφορες μελέτες, γιατί λοιπόν θέλει να αποσταθεροποιήσει ένα τομέα ο οποίος λειτουργεί καλά. Έχουμε αρκετούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πάνε καλά και που πρέπει να τους ασχοληθούμε, οπότε γιατί το 2007 πήραμε αυτά τα μέτρα που σίγουρα δεν είχαν αρκετά καλή βάση και να προχωράμε με αυτά. Δεν θα σας επαναλάβω τώρα όλα όσα ακούσαμε για αυτό το θέμα χτες, αλλά τώρα έχοντας ακούσει πολλούς επαγγελματίες, πολιτικούς, έχοντας διαβάσει και πολλές μελέτες για την προβληματική αυτή, Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποια συμπεράσματα. Μας είπαν πρέπει να ελευθερώσουμε τα δικαιώματα φύτευσης γιατί πρέπει να αυξηθεί το μέγεθος των επιχειρήσεων. Μα έχει αποδειχθεί από μια μελέτη ότι το μέγεθος της επιχείρησης δεν σημαίνει και οικονομίες κλίμακας και περισσότερες ε, ανταλλαγές. Μας είπανε ότι είναι πολύ ακριβά τα δικαιώματα φύτευσης. Ναι, αλλά έχει γίνει μια μελέτη που έχει δείξει ότι οι τιμές των δικαιωμάτων φύτευσης δεν επιβαρύνει σημαντικά ε, το κόστος δημιουργίας. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά γενικά αυτό ισχύει. Είναι επίσης σαφές ότι αν χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα φύτευσης με πολύ χαλαρό τρόπο και το είδαμε και στην Αργεντινή και στην ατικέν και στην πεδιάδα του Λούριου το είδαμε ότι δεν πλήττονται οι περιοχές. Είδαμε επίσης ότι η απουσία συστημάτων ρύθμισης φύτευσης στους ανταγωνιστές μας στις νέες χώρες δεν τους επέτρεψε να αποφύγουν ανισορροπία στις αγορές τους. Συνεπώς πιστεύω ότι το σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης τους επέτρεψε επέτρεψε στις περιοχές όπου υπάρχουν ε, αμπέλια να πάνε καλά. Υπάρχουν πολλά θετικά δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει καταρχήν να στηρίξουμε τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης με όλα τα καλά επιχειρήματα που γνωρίζουμε και που δεν θέλω να επαναλάβω πάλι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει από την άλλη μεριά ότι δεν έχουμε πρόβλημα μηχανισμού λειτουργίας των δικαιωμάτων φύτευσης. Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μεταφορές των δικαιωμάτων, με την εγκαθίδρυσή τους. Αν λοιπόν πούμε ότι καταρχήν θέλουμε να τα διατηρήσουμε, πρέπει από την άλλη μεριά να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλα αυτά τα προβληματικά σημεία, ώστε να έχουμε δικαιώματα φύτευσης σε όλες τις περιοχές και να αποτελούν ένα σύστημα ρύθμισης των αγορών που τόσο χρειαζόμαστε δεν έχει κανένα νόημα να θέλουμε να ανταγωνιστούμε τα φτηνά κρασιά των αναδυόμενων χωρών. Δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ με το δικό μας κόστος παραγωγής. Το μέλλον μας είναι η είναι ποιότητος. Και υπάρχει ζήτηση για τέτοια κρασιά ποιότητας είμαστε πάρα πολύ καλοί και στην εξαγωγή τους και στην κατανάλωσή τους. Αυτό είναι το μέλλον μας δηλαδή, είναι οι ποιότητες. Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι ναι, καταρχήν διατηρούμε τα δικαιώματα φύτευσης, αλλά είμαστε και έτοιμοι να συζητήσουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δομή, με το μηχανισμό, με την αποτελεσματικότητά τους και με την μεταφορά τους. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε άδικο όταν πρότεινε το μέτρο αυτό και πρέπει να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει το δόγμα της σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει. Γιατί ήδη έχουμε αρκετές χώρες, λείπουν νομίζω 30 ψήφοι για να έχουμε την ε, ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ο κύριος Τσόλος τη θέλει την πλειοψηφία αυτή πριν συμφωνήσει μαζί μας. Δικαίωμά του. Εγώ πάντα του λέω ότι η Κομοσιόν έχει το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας. Αν δεν θέλει να πάρει την πρωτοβουλία, θα την πάρουμε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε στη συναπόφαση τώρα. Και ο κύριος Νταντά είναι έτοιμος και πολλοί άλλοι από εμά να υποβάλουμε τις τροπολογίες που χρειάζεται για να αντιστραφεί το κλίμα και να μην έχουμε αυτήν την ακραία ελευθέρωση. Θέλουμε να χτίσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα φύτευσης το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και πάνω απ' όλα να αποφύγουμε κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές συνέπειες που δεν ξέρουμε καν πόσο θα μας στοιχήσουν. Εγώ πάντα λέω ότι δεν είναι η ΚΑΠ η οποία στοιχίζει ακριβά, η απουσία της να δείτε πόσο θα μας κόστιζε. Θα ήταν καταστροφικό να μην είχαμε τη ρύθμιση αυτή. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα συμφωνήσει με αυτά που παρουσίασα και εγώ αλλά και πριν από μένα ο κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Ο κύριος Αρντά έχει τώρα το λόγο. Α, η κυρία, η κυρία Αρντά διορθώνει ο πρόεδρος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, ονομάζομαι Ρομπέρτα Σαρντόνε. Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβολές σας. Νομίζω πως αυτό θα μας βοηθήσει στο να ολοκληρώσουμε καλύτερα την τελική μορφή της μελέτης μας. Θα προσπαθήσω να σταθώ σε κάποια ερωτήματα που τέθησαν. Όπως σας ε, ανέφερα, η διαδικασία απελευθέρωσης θα μπορούσε να συνοδεύεται από ένα κίνδυνο υπερπαραγωγής και επέκτασης της επιφάνειας που καλλιεργείται με κλίματα. Στην ουσία αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να ε, μας οδηγήσει στο να δούμε την παγκόσμια εξέλιξη των επιφανειών που καλλιεργούνται με κλίματα. Το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε μας λέει ότι σε περίπτωση απουσίας μελών ελέγχου του δυναμικού της παραγωγής, δηλαδή εάν γίνει κάτι όπως αυτό το οποίο γνώρισαν οι χώρες μη ε, εκτός ένωσης που δεν είχαν τον έλεγχο όπως έχουν οι δικές μας, ή τελικά τι γίνεται, διευρύνεται, επεκτείνονται οι επιφάνειες παραγωγής. Ε, εκεί όπου δεν υπάρχει έλεγχος, δηλαδή, οι επιφάνειες αντιδρούν στην ζήτηση της αγοράς. Εν τω μεταξύ όμως, η FDNA μας δείχνει ότι, μέσα σε μελέτη μας δείχνει ότι το, το επίπεδο Διατήρηση της καλλιέργειας των κλιμάτων ε, είναι μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες καλλιέργειες. Μπορεί δηλαδή να αυξηθεί η παραγωγή, ιδιαίτερα για εκείνους τους ε, παραγωγούς που θέλουν να στοχεύσουν σε ένα τμήμα της αγοράς με στόχο να ανταγωνιστούν με τους παραγωγούς εκτός Ένωσης στη διεθνή αγορά ε, παραγωγούς δηλαδή που μπορεί να ενδιαφέρονται στο να κάνουν μια παραγωγή σημαντική για τα κρασιά που εισήχθησαν με τη μεταρρύθμιση του 2008. Αυτά όσον αφορά την ανάλυση που έχουμε χρησιμοποιήσει και επίσης, και δεν το είπα στην παρουσίασή μου, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει απελευθέρωση, εμείς συστήνουμε να διατηρηθούν μέσα ε, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί τουλάχιστον ένα μίνιμουμ στάνταρ για τις επιφάνειες που μπορεί να καλλιεργούνται για παραγωγή ίνου ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα που είπατε, δηλαδή την μαζική μετακίνηση ε, επιφανειών από τις περιφερειακές, ε, από τις περιθωριακές, με συγχωρείτε, ε, περιοχές και να πάνε στην καλλιέργεια του, των αμπελιών σε πιο κεντρικές περιοχές. Ακόμα και με ένα προσωρινό μέσο ελέγχου, μετατράπηκε σε μόνιμο βέβαια κατά τη διάρκεια των ετών, όμως αυτό το μέσο δεν μπορεί να διαχειριστεί την ευελιξία την οποία χρειάζεται ο τομέας. Είναι απαραίτητο να ανανεωθούν οι κανόνες ε, των δικαιωμάτων φύτευσης. Αν τουλάχιστον αυτή η αναθεώρηση βοηθήσει στο να ξανασκεφτούμε αυτό το μέσο είναι καλό και είναι καλό που εστιάστηκε η προσοχή σε αυτή την αναθεώρηση την ε, μεταρρύθμιση. Τώρα, οι προβληματισμοί μας σε σχέση με την αλλαγή των ισχύων των, κανόνων ε, λειτουργίας για τη μεγαλύτερη διαφάνεια στο αγορά των ε, δικαιωμάτων προκύπτουν βασικά από μια ανάλυση που έγινε με βάση ένα ερωτηματολόγιο που διανύμαμε σε όλες τις χώρες παραγωγούς ίνου. Είχαμε συνεντεύχει στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ουγγαρία όπου ε, μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που μας οδήγησαν στο να τονίσουμε ότι υπάρχουν διαφορές στη λειτουργία ε, του τομέα και υπάρχουν επιτυχείς περιπτώσεις όπου όλοι είναι ικανοποιημένοι από τους μηχανισμούς λειτουργίας και αυτό συμβαίνει εκεί όπου η αγορά είναι διαφανής γιατί έχουν ήδη ας πούμε μηχανισμούς παρόμοιους με τους πληστηριασμούς και γι' αυτό υπάρχει και ένας μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο το δυναμικό παραγωγής και το, η ανταλλαγή των δικαιωμάτων φύτευσης δεν είναι το μόνο μέσο που διαχειρίζεται την παραγωγή παραγωγή, αλλά γίνεται η διαχείριση μέσω της συμμετοχής των ενώσεων παραγωγών και των επαγγελματιών του τομέα. Θα πρέπει δηλαδή να εμπνευστούμε από διάφορα πρότυπα ώστε να φτιάξουμε έναν μηχανισμό που να λειτουργεί με καινοτόμα, καινοτόμους κανόνες και με βάση τους γενικότερους κανόνες της ΚΑΠ. Και μια τελευταία παρατήρηση. Στην ανάλυση των στοιχείων της FADN προκύπτει ότι η διαχείριση των επιχειρήσεων έχει επιπτώσεις στο πιθανό κόστος της παραγωγής. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες οικονομίας κλίμακας στα κόστη παραγωγής. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο στοιχείο που θα πρέπει να καθορίσει τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής. Σίγουρα είναι ένα επιχείρημα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ο μοναδικός μηχανισμός που είναι σε θέση να ρυθμίσει την αύξηση του κόστου στο εσωτερικό του αμπελοϊνικού τομέα. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις λοιπόν, αλλά ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως ε, μάλλον τις τοποθετήσουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ελπίζω να απάντησα σε όλα τα ερωτήματα και σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις ε, που δώσατε. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης, που είναι η παρουσίαση της, από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας. ως ε, τμήμα της μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής και που εισάγει ε, νέα στοιχεία, νέα τεχνολογία ως μέσον για την γεωργία στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ξεκινήσει μια ε, εταιρική σχέση για την καινοτομία έτσι ώστε να προαγάγει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγή στον γεωργικό τομέα και τις χαμηλές εκπομπές. Αυτή η γεωργική εταιρική σχέση για την κοινοτομία μπορεί να επιτρέψει σε ενδιαφερομένους φορείς να συνεργαστούν ώστε να διευκολύνουν την εφαρμογή έρευνας και κοινοτομία σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές και η συνεργασία μπορούν να υποστηριχθούν από τον προτινόμενο κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η κυρία Βασίλια, εκ το λόγο παρακαλώ για να μας κάνει την παρουσίαση με μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο μιλητής χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε. Ο κύριος... Ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ε, δεδομένων των εξελίξεων στην ε, παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια της ε, υποχρέωσης να παράγουμε περισσότερα για λιγότερο, κόστος, να σας παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ε, καινοτομία με την ε, πρόταση της 29 Φεβρουαρίου και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 γιατί αυτή η ΕΣΚ, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας θα πρέπει να αποτελέσει ένα μέσον εξυπηρέτηση των στόχων μας και μάλιστα σε ένα δεδομένο, με δεδομένο το ε, κλίμα της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Ποια είναι τα ζητήματα λοιπόν που θα να επιλύσουμε. Καταρχάς την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα 70% για 2050 ε, όπως μας λέει η Διεθνής η Οργανώση Τροφίμων και Γεωργίας and Agricultural Organization που σημαίνει η δημογραφική δηλαδή αύξηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ σημαντική έκρηξη στη ζήτηση τροφίμων ε, γεωργικών προϊόντων δηλαδή στον κόσμο και άλλη γεωργική παραγωγή θα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο παρελθόν το κέρδος παραγωγικότητας ε, που εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Γεωργία ανερχόταν σε 20% ανά δεκαετία. Τέτοιο κέρδος όμως παραγωγικότητας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο επί τη βάση των υφισταμένων τεχνολογιών και θα πρέπει συμπληρωματικά να ε, συμπληρωθεί αυτό το κέρδος παραγωγικότητας με την αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των αρνητικών συνεπειών αυτών στο περιβάλλον. Κύρια πρόκληση της ε, γεωργίας για τις επόμενες δεκαετίες, οι δεκαετίες θα είναι ως εκ τούτου η παραγωγή περισσότερων με λιγότερο κόστος, δηλαδή more with less, δηλαδή μια μετατόπιση των στόχων και του ε, τρόπου επίτευξη των στόχων. Άρα χρειαζόμαστε καινοτομία έρευνα σε κάθε τομέα προσαρμοσμένη σε νευρή φάσμα δομών και αναπτύξεων και από την άλλη πολλοί ήταν οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι υπογραμμίσαν ότι υπάρχει κίνδυνος ε, συμφόρησης όσον αφορά την καινοτομία στη γεωργία δηλαδή απουσία σχετισμού μεταξύ γεωργικής έρευνας αφενός και γεωργικής πρακτικής αφετέρου. Η καινοτομία λοιπόν, η εταιρική σχέση για την καινοτομία στη γεωργία και τη βιωσιμότητα θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της προκειμένου. Και θα ήθελα να ε, προτείνω την ενίσχυση και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρηματικών, γεωργών, επιστημόνων, ακαδημανικών κύκλων, διοικητικών φορέων που θα επιτρέπουν την ε, ταχύτερη διαβίβαση της πληροφορίας από την επιστήμη στην ε, πράξη και που θα εξασφαλίζουν ταυτόχρονα η ε, ικανοποίηση των αναγκών με βάση τα στοιχεία που θα προσφέρει η επιστημονική κοινότητα. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν μπορεί να αποτελέσει, να διαδραματίσει ρόλο καταλητικό και να στηρίξει μέσα και δομές χωρίς να τα επαναλάβει, χωρίς, να, χωρίς τις επικαλύψεις δηλαδή. Αυτή θα είναι η δύναμη της, αυτή θα είναι η προσθέμενη αξία ενώ η πολιτική για την ανάπτυξη πέθρου μέσα σε μαζί με ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την ε, καινοτομία, την έρευνα και την καινοτομία θα μπορούν να αποτελέσουν τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές, πολιτικές πάνω στις οποίες θα στηρίζεται η ΕΣΚ για να υποστηρίξει τις καινοτόμες δράσεις. of the EAP. Οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Θα αξιοποιήσουν μέτρα λοιπόν καινοτομία για την πολιτική του, για την ανάπτυξη πέθρου, ιδιαίτερα με την ενεργοποίηση διαφορών ομάδων δράσεω ή λειτουργία, ε, διάδοση των πληροφοριών, διάδοση επίση των ε, λύσεων για τρόφιμα, κύρια μέτρα Ε, θα έχουν να κάνουν με τα φυσιολογικά ή ε, γεωγραφικά δεδομένα, επιστημονικά στοιχεία και άλλες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η καινοτομία και η τεχνολογία. Με βάση την καινοτόμο δράση επιτόπου. Κυρίες δράσεις μπορούν να αποτελέσουν ε, προγράμματα εφαρμοσμένα πολυτομεακές προσεγγίσεις και υποστήριξη στην καινοτομία. Δύο πολιτικές συμπληρωματικές που ενισχύουν η μία την άλλη. Οι δράσεις των προγραμμάτων ανάπτυξη πέθρου εν γέννη εφαρμόζονται στο πλαίσιο κάποιων περιφερειών ε, προγραμματισμού, ενώ η ερευνητική πολιτική ξεπερνά την κλίμακα αυτή. Και συγχρηματοδοτεί καινοτόμε δράσεις και βεβαίως περιφερειακά, διασυνοριακά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ όλων των φορέων, για να συγκεράσουμε τις προσπάθειες της επιστήμης με αυτές τις πράξεις, έχει προταθεί θέσπιση ενό δικτύου επικεντρωμένου στην καινοτομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποτελεί την ψυχή της ΕΣΚ και που θα ενθαρρύνει ομάδες λειτουργίες ε, θα, θα τις στηρίζει στις βάσεις δεδομένων τους, θα τους προσφέρει προτάσεις. Επίσης θα έχουμε την ομάδα, διευθυντική ομάδα υψηλού επίπεδου που στο στόχο θα έχει να εξασφαλίσει την ε, απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, δηλαδή δεν θα έχει ε, εξουσία για λήψη αποφάσεων, απλώς θα θέτει σε εκείνη τη διαδικασία και θα ε, δίνει κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία μέσα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου. Η διακυβέρνηση της ΕΣΚ θα εξαρτάται από τις υφιστάμενες δομές, όπως άλλωστε ανέφερα νωρίτερα. Το περιεχόμενο και οι προτεραιότητες που θα ε, επιδιώκει να εξυπηρετήσει η ΕΣΚ θα αφορούν δραστηριότητες όπως γεωργική δραστηριότητα, διαχείριση φυσικών πόρων, στήριξη υπηρεσιών οικοσυστήματος, υποστήριξη της ασφάλειας σε προμήθεια τροφίμων και Κλείνοντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη πως η ΕΣΚ για την γεωργία έχει σημαντικό δυναμικό να προσφέρει και μπορεί να συμβάλλει στον στόχο μιας ε, ανάπτυξης, όπως την ορίζει η στρατηγική του 2020, ε, εφιούς και βιώσιμης. Ζητάει βέβαια η Επιτροπή την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων φορέων για την ε, υλοποίηση και την εφαρμογή αυτού νέου μέσου και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλό σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει να αποδεχθεί την θέση λειτουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Κοινοτομία όπως την περιγράφει η ανακοίνωση της 29 Φεβρουαρίου. Φυσικά όλα αυτά με κάθε επιφύλαξη των ακόμη εκκρεμών ζητημάτων σε επίπεδο Επιτροπής όπως μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής που σχετίζονται σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Οικονοτομία. Με στόχο πάντα να θεσπιστούν τα το απαραίτητο πλαίσιο και δικτύωση ε, με την ε, ε, διευθυντική ομάδα με το Διευθυντικό Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου που θα προσδιορίζει ένα στρατηγικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει το, τα της σύνθεσης αυτού του ε, δι, Διευθυντικού Συμβουλίου και εν αυτό το χρόνο θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο ζητώντα τη συμμετοχή του σε αυτό. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Συζήτηση τώρα. Η κυρία Ρέιμερς πρώτη που θέλει το λόγο. Äh, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την παρουσίαση της σύμπραξης ε, για την κοινοτομία. Είναι σωστό βέβαια να υπάρξει ένα δίκτυο που θα εξασφαλίζει την ανταλλαγή, την επικοινωνία μεταξύ αυτό που ασχολούνται με την έρευνα βάσης και εκείνων που βρίσκονται στο πεδίο, στην εφαρμογή. Πολλές φορές στο παρελθόν είχαμε δηλαδή αποτελέσματα έρευνας που δεν ήταν ε, δυνατόν να, μετατραπούν σε πράξη, δεν μπορούσαν να μεταφραστούν σε πρακτικά αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να είναι η επιδίωξή μας λοιπόν, να προχωρήσουμε ταχύτερα στην εφαρμογή της έρευνας. διότι νομίζω ότι πολλές φορές ε, όταν ε, τίθεται ζήτημα να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα, ίσως να επικρατεί σύγχυση σε επίπεδο είτε της κοινότητας των επιστημόνων, είτε της κοινότητας που ασχολείται με την εφαρμογή στην πράξη αυτού του αξιώματος και άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ πρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσίαση. Δεν θα το σαφή για μένα τα πράγματα. Θα ήταν καλό να το δούμε γραπτό για να καταλάβουμε τι μορφή ακριβώς προβλέπεται να λάβει. Διότι μας φαίνεται πολύ θεωρητική όλη αυτή η προσέγγιση και θα πρέπει να δούμε στην πράξη εάν υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένες ε, ερευνητικές ε, κατευθύνσεις, συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς να τους προχωρήσουμε μέχρι την πρακτική εφαρμογή. Γιατί για ορισμένου μπορεί να έχουμε φερειπίν επιφυλάξει όπω γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Ή μπορεί σε άλλου να θέλουμε να δώσουμε προσθεριώθηση, όπω την έρευνα για την προστασία του περιβάλλοντο μέσα από τη γεωργία, στην οποία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Επίση, λέ, λέγεται ότι η FAO έχει πει ότι πρέπει να παράγουμε 70% περισσότερο. Όχι, δεν το έχει πει αυτό η FAO. Τουλάχιστον έχει με αυτού του όρου. Απλώς μας λέει ότι αν δεν αλλάξει τίποτα στον τρόπο παραγωγής θα χρειαστεί να παράγουμε 70% περισσότερο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα παράγουμε, θα χρειαστούμε να παράγουμε 70% ε, περισσότερο και αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο είναι καλό να μην διαδίδεται τόσο εύκολα. Βεβαίω η παραγωγή μα πρέπει να γίνει πιο βιώσιμη. Βεβαίω κάποιε από τι λύσει στι οποίε αναφερθήκατε είναι σωστέ. Δηλαδή η πραγματική πρόκληση είναι να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα πράγματα, με λιγότερου πόρου. Αλλά το βασικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το σύστημα όπως έχει τώρα δεν, δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κύριε Μαγκίνες, παρακαλώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την περίμενα την παρουσίαση αυτή γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που προσπαθούμε και είναι σαν να ανακαλύπτουμε εκ νέου τον τροχό φαίνεται να λειτουργεί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το μοντέλο μπορεί να ξανακάνει τη δουλειά που πρέπει. Έχω βέβαια κάποιες αφιβολίες επειδή πρόκειται για ακαδημαϊκή μελέτη, αλλά νομίζω ότι είναι σωστή η ιδέα. Ότι είναι καλό να έχουμε καλή έρευνα σε καλό επίπεδο, απλώς ακόμα δεν ξέρω πώς θα το πετύχουμε. Δεν μιλήσαμε για τον προπολογισμό, δεν μιλήσαμε για τέτοια πράγματα, δεν ξέρω αν προβλέπονται. Η εμπειρία μας από την εταιρική σχέση σε θέματα καινοτομία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να το διευκρινίσει ίσως περισσότερο. Έχουμε πάρει κανένα μάθημα από αντίστοιχες προσπάθειες στο παρελθόν. Πάντως αυτή η πρωτοβουλία ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το έχουμε πει ξανά και ξανά στην Επιτροπή μας και θα το λέμε ξανά και ξανά. Το θέμα είναι ότι πώς θα φτάσουμε ε, στο επίπεδο του... της γεωργικής ε, γης. Φυσικά και το θέλουμε και διψάμε για γνώση. Σίγουρα θα βοηθήσει. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει άλλος κανείς το λόγο. Παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τις προτάσεις που ακούστηκαν. Πραγματικά, η ιδέα να ξεκινήσει η ανακοίνωση αυτή έτυχε θετικής αποδοχής. Έτσι κι Μιλάμε για βιωσιμότητα εδώ, όχι για παραγωγικότητα, αλλά για βιωσιμότητα. Άρα λοιπόν ο στόχος δεν είναι μόνο αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά να διασφαλίσουμε επίσης ότι θα είναι και βιώσιμη αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας. Αναφερθήκαμε στο, στη δυνατότητα του 70%. Βέβαια παραμένει μια υπόθεση. Ακόμα όμως και αν δεν είναι ο ακριβής αριθμός, ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση στη ζήτηση και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να τη στηρίξει. Αυτός είναι και ένας ε, από τους στόχους της προσέγγισης αυτής. για την ε, βιολογική παραγωγή και την παραγωγή ποιότητας θα έχουμε άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για τα νέα αυτά μέσα. Έρχομαι τώρα στο θέμα του προπολογισμού. Δεν χρειάζεται να έχουμε έναν ειδικό προπολογισμό γιατί η πρωτοβουλία αυτή κατευθύνεται στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σχέση ανάμεσα στους ερευνητές, τους συμβούλους, τους ενδιαφερόμενους, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τη μία και τους ε, γεωργούς από την άλλη. Έτσι ώστε η γνώση να περάσει από τους ερευνητές ε, στους γεωργούς. Και από την άλλη μεριά να υπάρξει και feedback όμως από τους παραγωγούς προς τους ερευνητές. Αυτό είναι ο κύριος στόχος της ιδέας αυτής. Ο προπολογισμό βέβαια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά όταν έχουν αναπτυχθεί περισσότερο τα προγράμματα για το λειτουργικό στάδιο. Προβλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί κάτι στα πλαίσια αυτής της νέας ιδέας από κάτω προς τα πάνω, bottom-up. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν πρέπει να πω ότι δεν είναι ακαδημαϊκής φύσεως αυτό που κάνουμε γιατί δεν σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε σε νέα έρευνα αλλά να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ήδη υπάρχουσα γνώση και να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι αγρότες και οι ερευνητές. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια νέα ακαδημαϊκή προσέγγιση όπου θα χρειαστεί νέα τεχνολογία, θα υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και επενδύσεις για κάποια νέα προγράμματα. Η προσέγγιση δεν είναι ακαδημαϊκής φύσεως, λοιπόν. Εμείς θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ελαστικοί. Γι' αυτό εξάλλου και ζητήσαμε από όλους τους ε, εταίρους μας στο Κοινοβούλιο να μας βοηθήσουν να χτίσουμε καλύτερα την ιδέα αυτή. Και γι' αυτό και υπάρχει και αυτό το steering board, μια διευθύνουσα, ένα διευθύνων σώμα, το οποίο θα βοηθήσει περισσότερο να αναπτυχθεί αυτή η ιδέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τώρα. Που είναι το σημείο 17. Ορισμός εισηγητών. Α, δεν έχουμε τίποτα σήμερα. Από αυτό. Ωραία. Επόμενο σημείο. Η επόμενη προσεχή συνεδρίαση. Προσεχή συνεδρίαση 27 Μαρτίου 2012. Στις 3. Τρίτη. 27 Μαρτίου λοιπόν. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους. Meeting of the Committee of Agriculture. Thank you very much. Thank you. Thank you for interpreters and for, for all.